Πρέπει να ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Έχει πάει 3 και τέταρτο και πρέπει να ξεκινήσουμε. Το πρώτο θέμα μας σήμερα είναι η έγκριση φυσικά των πρακτικών. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε επίσης και την παρουσίαση της μελέτης από εξωτερικούς συμβούλους για την πρωτοβουλία των πολιτών. Έχουμε επίσης και εκθέσεις για την πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τις έκθεσης για την αποστολή μας στην Ελλάδα. Αύριο το πρωί θα έχουμε επίσης και μια μεγάλη συζήτηση 30 αναφορές σχετικά με την προστασία των παιδιών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δανία. Η ημερήσια διάταξη σήμερα θα γίνει σεβαστή εκτός από το σημείο 8 γιατί ο κύριος Higgins μου ζήτησε να αναβάλουμε το θέμα του γιατί δεν θα είναι παρόν. Για το σημείο 8 λοιπόν αναβάλλεται η συζήτηση. Όταν θα είναι παρόν θα τεθεί το θέμα. Θα έχουμε επίσης και αναφέροντες για 5, 8, 16 και 15. Θα έχουμε παρουσία εμπειρογνωμόνων για το 9 και για το 14 θα έχουμε και εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, τον κύριο Λιώκα, αν ακούσαμε το όνομα καλά και θα κάνει μία δήλωση στην Επιτροπή μετά από την αυριανή ψηφοφορία. Δεν έχω κάτι άλλο να σας παρουσιάσω. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο στην σημερινή διάταξη. Ο Βαλένζα, ευχαριστώ Πρόεδρε, στο σημείο 2 στην έγκριση των πρακτικών του μηνός Δεκεμβρίου. So, everybody... Λοιπόν, όλοι συμφωνήσατε για τα πρώτα θέματα. Γίνεται δεκτή λοιπόν η μερίσια διάταξη. Το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών. Της 16ης Δεκεμβρίου εδώ κύριε Βαλέντσα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επαναλαμβάνω να αναβληθεί η έγκριση των πρακτικών. Αυτό θα ήταν σωστό γιατί σύμφωνα με τον κύριο Ήτου Γκάιζ υπάρχει λάθος κάπου στα πρακτικά αυτά. Δεν ξέρω λεπτομέρειες τώρα σχετικά με το θέμα, αλλά καλό θα ήταν να το αναβάλουμε μέχρι ότου έχουμε κάποιες διευκρινήσεις. Ο κύριος Ίτογκάης θα το εκτιμήσει δεόντως. Κύριε Τσίτσεστερ και τα υπόλοιπα μέλη, συμφωνείτε με το αίτημα του κυρίου Βαλένζα να αναβληθεί δηλαδή η έγκριση του υπαριθμών δύο θέματος. Καλώς στις 16 Δεκεμβρίου λοιπόν αναβάλλεται το τρίτο θέμα ως συνήθως έχουν διανεμηθεί τα έγγραφα και δεν έχουν ληφθεί σχόλια για τις συστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται και θεωρούνται πλέον δεκτές. Περνάμε τώρα στην πρώτη αναφορά. Πρόκειται για την αναφορά που κατέθεσε η κυρία Άννα Κλέτς της Πολωνίας, από την Πολωνία. Είναι παρούσα η κυρία Κλέτς και θα της δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την υποστήριξη της αναφοράς μου και τη δυνατότητα που έχω να έρθω να μιλήσω. Εκπροσωπώ μία οργάνωση που αναπτύσσει προσπάθειε προσπάθειες της 15 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από ό,τι μαθαίνουμε Υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα και πρέπει να συζητηθεί ε, το θέμα της παρηγορητικής αγωγής στις διαφορές χώρες. Ιδιαίτερα για την Ιταλία θα γίνει αναφορά από ό,τι μαθαίνω στην ημερήσια διάταξή σας και προβλέπετε. Πάντως ε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση που αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται για λόγους χρόνιας ασθενείας είτε στο σπίτι είτε στο νοσοκομείο κατάκητοι. Εγώ δεν είμαι γιατρός, είμαι απλώς ασθενής και θέλω να εκπροσωπήσω με τη φωνή μου εκείνους οι οποίοι υποφέρουν από πολύ βαρύς πόνους. Ε, από την εμπειρία μου διαπιστώνω ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για την αντιμετώπιση του πόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσο δύσκολες συνθήκες, πολλοί ασθενείς πολλές φορές διαπράττουν, ε, φτάνουν ακόμη και μέχρι την αυτοκτονία γιατί δεν αντέχουν τους πόνους. Είναι λοιπόν άξιο απορία το πώς μπορούν στον 21ο αιώνα να παραμένουν χωρίς την κατάλληλη παρηγορητική αγωγή, χωρίς τα κατάλληλα αναλγητικά, τόσοι πολλοί άνθρωποι. Ενώ το 2013 διαπίστωσαν τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν προσφέρονται ε, ότι όταν δεν προσφέρονται αναλγητικά στον ασθενή αυτό μπορεί να αποτελεί να αναγνωριστεί και ως μορφή βασανιστηρίου και άρα παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φροντίσετε για την θέσπιση ενιαίων κριτηρίων για την παροχή αναλγητικών φαρμάκων, για την παρηγορητική αγωγή. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον κάθε έναν μας, την κάθε μία μας και εσάς όσο και εμένα και όλους τους συγγενείς ή γνωστούς μας. Γι' αυτό λοιπόν να στεθεί πλέον ένα τέλος στην αδικία αυτή που διαπιστώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αναφερθώ και σε στατιστικά δεδομένα, το 2013 χορηγούνταν 413 μιλιγκράμμ αναλγητικών ε, στην ε, Γερμανία κατά ασθενή, στις ΗΠΑ 648 μιλιγκράμμ για την ίδια περίοδο και στην Πολωνία μόνο 40 Πέντε. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία, ότι έχουμε πολύ χαμηλότερα ποσοστά ε, κάλυψης ε, από οποιούχα αναλγητικά στην Πολωνία ε, με το επιχείρημα ότι μπορεί να προξενήσουν εξάρτηση οι γιατροί δεν τα χορηγούν στους ασθενείς ενώ υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να διατεθούν υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί που ασχολούνται με την παρηγορητική αγωγή και πολλά μέσα που διαθέτουμε για την υποστήριξη των ασθενών. Υπάρχουν ε, έρευνες ε, του 2010 αλλά και μεταγενέστερες, ακαδημαϊκές δηλαδή εργασίες ε, που αναπτύσσονται σε διάφορα ερευνητικά κέντρα και που παράγουν συστάσεις για τα κράτη-μέλη. Και οι οποίες έχουν σαν αντικείμενο την ε, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για τα φάρμακα αυτά. Ωστόσο τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιήθηκαν στην εν έρευνα είναι αρκετά παλιά, του 2002 τα δεδομένα τα οποία αξιοποίησαν οι Πολωνοί ερευνητές και έτσι δεν έχουν καμία επικαιρότητα, δεν είναι σύγχρονα και δεν μπορούν να είναι αξιόπιστα. Σε αυτό οφείλεται και η άνηση πρόσβαση στα αναλγητικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να εκτιμήσει πόσο πονάει ο ασθενής. Αλλά έχουμε να κάνουμε με μία πτυχή και οικονομική η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρώπη ασφαλώς μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Έχουμε να κάνουμε τεράστια ποσά και γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει κοινά κριτήρια και προδιαγραφές για τη χορήγηση αναλυτικών σε όλους τους ασθενείς για να υποστηρίξουμε τους ίδιους ασθενείς αλλά και τους οικείους τους. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των ασθενών και των ε, οικογένειών τους. Ευχαριστώ και είμαι σε θέση σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βέρνερ από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αναφερομένη, λαμβάνω το λόγο εδώ έχοντας διαβάσει την αναφορά σας προσεκτικά και στις λεπτομέρειες και μπορούμε σε ένα βαθμό να δώσουμε ε, το πράσινο φως στην αναφορά σας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα βαθμό. Όπως είπατε ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητα αποκλειστική στην υπόθεση αυτή, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να διατυπώσουμε κατευθυντήριες γραμμές, εφαρμόσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Κατά την έποψή μας θα ήταν καλύτερο να ενθαρρυνθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η Pain Alliance Europe, να συντάξουν κατευθυντήρες γραμμές οι ίδιες και να εξασφαλίσουν συμφωνίες με εθνικές οργανώσεις και φορείς στον τομέα αυτών. Φυσικά η Επιτροπή είναι διτεθειμένη να υποστηρίξει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με ε, διάθεση ενδεχομένως πηγών και ενημέρωση για κατευθυντηρίες γραμμές που ισχύουν σε κράτη-μέλη, σε μια προσπάθεια υποστήριξη συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και βεβαίως θα ήμασταν διατεθειμένοι εφόσον αυτό μπορεί να εγγραφεί στο ετήσιο πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να χρηματοδοτήσουμε με το δικό μας προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία ε, έργα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του πόνου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ για την διαθεσιμότητά σας. Ο κύριος Βαρέντσα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να αναλάβουμε μέτρα για να διατυπώσουμε κοινέ κοινές προδιαγραφές, κοινά κριτήρια. Τα όσα ακούω από την Επιτροπή δεν με ικανοποιούν σαν απάντηση και γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την υπόθεση αυτή. Ίσως να είναι δυνατή η συλλογή του ενός εκατομμυρίου υπογραφών, οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο οφείλει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αναφέρθηκε σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Βεβαίως μπορούν και αυτές να συμπράξουν και πιστεύω ότι μπορούμε από κοινού να εξασφαλίσουμε την ε, ενασχόληση της Επιτροπής με τα προβλήματα αυτά που μας αναφέρατε. Παρακαλώ κύριε Μπαλντίνη. Ε, ε, ναι, ευχαριστώ. Έχω το κείμενο της Λίδια Γκέριγκερ και θα σα το διαβάσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχά να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορούσα σήμερα να είμαι παρούσα και προσωπικώ εκφράζω την στήριξή μου στην αναφορά αυτή. Η αναφορά της κυρίας Ανακλές για την εισαγωγή ενιαίων διαδικασιών στην Ευρώπη για την αγωγή και τη θεραπεία του μακροχρόνιου πόνου είναι πολύ σημαντική. Μας εξηγεί η αναφέρουσα τις ε, δραματικές προσπάθειες που κατέβαλε μέσω της ασθένειας και τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί στην Πολωνία αρνήθηκαν να τις χορηγήσουν ε, ε, καταπραϊντικά ενεργητικά φάρμακα για να αντιμετωπίσει τον απίστευτο πόνο που αισθανόταν. στην Πολωνία αποτυπώνεται αυτό μέσω της χρήσης της ε, μορφήνης που είναι 10 φορές χαμηλότερη από τη, από τη... από Γερμανία. Και υπάρχει άρνηση χορήγησης ε, αναλγητικών ε, προς ασθενείς και το οποίο θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι είναι ένα είδος μαρτυρίου. Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να δούμε ποιε είναι οι αιτίε αυτή τη τάση. Κατά πόσον είναι ένας τρόπος περικοπής κόστους ε, για τα νοσοκομεία, ένα πρόβλημα πρόσβασης ε, στα φάρμακα ή ε, η ανησυχία ότι η ασθενείς μπορεί απέναντι στην ε, αγωγή τέτοιων φαρμάκων Θα ήθελα λοιπόν να εισηγηθώ την ε, θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων για τη χορήγηση τέτοιων φαρμάκων και την, ε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, η Λίδια Γκέρινγκερ de Ödenberg. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει πρόεδρος. Να ρωτήσω το εξής τον κύριο Βέρνερ. Δεν μου είναι σαφές για ποιον λόγο η Κομισιόν δεν μπορεί να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές ε, στην περιοχή αυτή. Γιατί η Επιτροπή δεν θα μπορούσε να προβλέψει μια ομοιόμορφη, ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία για την αγωγή ε, μακροχρόνιου, χρονίου, πόνου. Και ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα. Γιατί να δίδονται πόροι σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις αφενός, αλλά αφετέρου να μην μπορούν να θεσπιστούν κάποιες ε, κοινέ κατευθύνες γραμμές. Πρόεδρε, ευχαριστώ, λέει ο κ. Βέρνερ. Αν μιλούμε για κατευθυντήρες γραμμές που θα υιοθετούσε η Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προβλέπεται μια διαδικασία. Αυτό κυρίως λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με την συνθήκη ο ορισμός των πολιτικών υγείας και η οργάνωση και η χορήγηση θεραπείας και φαρμάκων είναι υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν θα συμφωνούσαν προς την θέσπιση μιας διαδικασίας που θα προέβλεπε κατευθυντήρες γραμμές στην περιοχή αυτή αρμοδιότητάς τους. Και γι' αυτό προσεγγίζουμε με γενικό τρόπο αυτές τις χρόνιες ασθένειες και ειδικά το θέμα της αντιμετώπισης του πόνου συνεργαζόμενοι με μη κάπα όμικρον και χρηματοδοτώντας έργα την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών στην περιοχή μέσω του προγράμματος υγείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι ευρωπαϊκές κατευθυντήρε γραμμές, σημαίνει απλώς ότι αυτές όλες οι οργανώσεις, όλοι αυτοί οι φορεί στην Ευρώπη θα μπορούσαν να φτάσουν σε μια συμφωνία με όλους τους υποκείμενους φορείς και οργανώσεις ώστε να υπάρξει μια όθηση, μια πολιτική όθηση ώστε οι κυβερνήσει των κρατών μελών να εφαρμόσουν να ζητήσουν δηλαδή την εφαρμογή αυτών που θα έχουν συμφωνηθεί σε αυτές τις κατευθύνες γραμμές. Προτείνω να αφήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή και να ζητήσουμε κάποιες definitions, γιατί νομίζω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν, οπότε θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα ζητήσουμε περισσότερες διευκρινήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές και την υιοθέτηση γενικότερων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή. Θα επανέλθουμε στο θέμα αργότερα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι. Έχετε ένα λεπτό για να απαντήσετε, να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλω να πω ότι εδώ τα, η παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων των ασθενών δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτε άλλο από μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί και ο ασθενή άνθρωπο είναι. Και αν του στερήσουμε την πρόσβαση στο αναλγητικό, στο φάρμακο, τότε τον βασανίζουμε. Άρα έχουμε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Thank you again. So we Ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα θα περάσουμε στην επόμενη. So we have another change because... Υπάρχει μια μικρή αλλαγή γιατί όπως είπα ζητήθηκε αναβολή της 6 οπότε θα περάσουμε αμέσως στην 7 αναφορά του Στέφανο Τζοβανίνη Ιταλού για την εξαίρεση από την Οδηγία 2006 σχετικά με τον εκ των παραχωρήσεων των θαλάσσιων χώρων από το Ιταλικό κράτος. Θα του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης και τους ε, μαθητές από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας της Ατσέρα οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τη συνεδρίασή μας. Η Επιτροπή μας γνωρίζει καλά τον Δήμο της Ατσέρα. Είχαν έρθει εκπρόσωποι της πόλης αυτής ε, όταν ε, είχε τεθεί το θέμα των αποβλήτων. Με την παρουσίαση αυτή θέλουμε να τονίσουμε ε, κάποιες πτυχές ε, σχετικά με τις παραχωρήσεις ε, ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Χρειάζεται μεγαλύτερη εμβάθυνση. Στην απάντηση της Κομισιόν υπάρχει, λέγει η Κομισιόν ότι το άρθρο 12 της Οδηγίας Υπηρεσιών αναφέρεται στους φυσικούς πόρους. Εάν εξετάσει κανείς το άρθρο 12 δεν επιτρέπεται αυτή η ερμηνεία, διότι αυτή η έννοια είναι αρκετά ασαφής και δεδομένης Δεδομένου των συνεπειών μια τέτοια ασάφεια ερμηνεία, χρειάζεται να εμβαθύνουμε και να εξετάσουμε δελεχέστερα ποιοι είναι εκείνοι οι φυσικοί πόροι που έχουν αντίκτυπο και που θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο ε, περιοριστικού καθεστώτος. Και ποια, ποιοι είναι οι φυσικοί πόροι που τους, το, θεωρεί το Ιταλικό κράτος εκμεταλλεύσει τους πόρους. σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία του τριτογενού, των υπηρεσιών ε, τριτογενού και την παροχή των υπηρεσιών τριτογενού τομέα. Για τις ε, ε, περιοχές και τις παραλίες θεωρούμε ότι δεν εμπίπτει στον περιοριστικό αυτό ε, ορισμό η, η θεώρηση της Κομισιόν, αλλά σε φυσικό πόρο ε, σπάνιο θεωρώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιβεβαιώσει την σπανιότητα του φυσικού αυτού πόρου, αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Και παραθέτω κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό. Προερχόμενο από ένα έγγραφο του Υπουργείου Αιγείας από το 2010, η Ιταλία έχει τον 4.421 ε, παραλίες που είναι ο υψηλότερος αριθμός στην Ευρώπη 35,8% του συνόλου των ε, παραλιών της Ευρωπαϊκής Υπήρου, λέει ο μιλτής. Προκύπτουν αυτά από, ένα, από δεδομένα του 2011. Έχουμε περίπου 5.000 χιλιόμετρα από το σύνολο των ακτών που χρησιμοποιούνται για παραλίες. Ένα 18% εξ αυτών είναι αντικείμενο παραχωρήσεων. Άλλο ενδιαφέρον δεδομένο από 2.000 έχουν διπλασια... που ήταν το 2011 έχουν διπλασιαστεί. Δηλαδή έχουμε νέες παραχωρήσεις κάθε χρόνο χωρίς αποκλεισμό επί τη βάση εθνικής ε, υποβολής και, το, και χωρίς πλήρη εξέταση των εγγράφων των υποβολών που γίνονται σχετικά με τις παραχωρήσεις αυτές. Ε, η Ισπανία μέσω πρόσφατης νομοθεσίας μπόρεσε να μεταρρυθμίσει ε, τη νομοθεσία που διέπει τις, ε, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και τις παραχωρήσεις που αφορούν σε ακίνητα και σε ε, περιοχές. Μεταξύ των παραχωρήσεων θαλασσίων χώρων έχουμε ξενοδοχειακέ εγκαταστάσει, πάρα πολλά εστιατόρια ο μιλητής αναφέρει με τεράστια ταχύτητα και η κυρία Βίβιαν Redding, Επίτροπος ε, Δικαιοσύνης, ε, συνεχάρει τον Ισπανό ε, Υπουργό για, τον, για την πρωτοβουλία αυτή, ώστε να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι όταν μιλούμε για την το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου περιουσιακού στοιχείου. Στην η Ιταλία αναρωτιέμαι αντιστοιχεί, ανήκει στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκει η Ισπανία. Και όταν μιλούμε για εξαιρέσεις τριακονταετία, αυτό το υποστήριξε στεναρά και η Επιτροπή εσωτερική ε, εγχώρια οικονομία, χωρί όμω να λάβει υπόψη τη την συνολικότερη εικόνα της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των παραλίων στην Ευρώπη θεωρούμε ότι αυτές οι παραχωρήσεις όχι μόνο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αλλά πρέπει να δούμε και κατά πόσον κοινωνικός και οικονομικός αυτές οι επιλογές είναι οι ορθές επιλογές. Σε σχέση με, τις, με τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν και σε σχέση με το, τυχόν θετικό ε, ε, οικονομικό όφελο ή αντιστάθμισμα. Αυτή τη στιγμή οι δικαιούχοι των παραχωρήσεων είναι υπήκοοι διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο Ιταλοί και μεταξύ των προϋποθέσεων που υποτίθεται ότι επιτρέπουν την ανάπτυξη του συστήματός μας συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες κατευθύνονται προς τη χρεοκοπία και είναι δηλαδή ανασφαλής οικονομικά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα μια πλήρη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της το σύνολο της Ιταλικής νομοθεσίας, την ελευθερία ε, μετακίνησης ε, και παροχής υπηρεσιών, αλλά και περιβαλλοντικές ε, και οικονομικές πτυχές. Θα ζητούσα λοιπόν και πολιτικός να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ενδελεχέστερα την όλη αυτή διαδικασία μέσω των τοπικών αρχών εκπροσώπησής μας και διαφημίζοντας ότι η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε εξαίρεση υπό το άρθρο 37 σχετικά με τη μετανάστευση. Δεν υπήρξε λοιπόν ο χρόνος ε, ώστε να εξεταστεί πλήρως η συμβατότητά του με τις Ευρωπαϊκές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ το λόγο για την αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα εμείνω στα τρία στοιχεία τα οποία έθεσε ο αναφέρον. Καταρχάς το θέμα των φυσικών πόρων. Δεν σταθήκαμε στην επιστροφή που δώσαμε, στην επιστροφή στο άρθρο 12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει πάντως ότι όταν μιλάμε για περιορισμένους φυσικούς πόρους ή σπάνιδα φυσικών πόρων, όπως λέγει το άρθρο 12, πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν πόροι φυσικοί και αναφερθήκαμε στις ακτές εδώ και το κράτος είναι ιδιοκτήτης και για τις οποίες αυτές περιοχές σε κάποια φάση απαιτείται μια κάποια με διαφανή και ανταγωνιστικό τρόπο εκμετάλλευσή τους. Ε, το ότι μιλήσαμε λοιπόν για περιορισμένους πόρους και όχι για σπάνιδα πόρων, αυτό δεν, αφορά, δεν δημιουργεί κάποια δυσκολία. Σχετικά με το θέμα ακριβώς της σπανιότητας αυτής το ότι πρόκειται για παραλίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφεαυτού είναι ένας πόρος περιορισμένος. Περιορισμένος όχι μόνο γιατί ε, δεν υπάρχει παρά ένα συγκεκριμένο ε, έδαφος ε, παράκτιο στο οποίο αναφέρεται και ο συγκεκριμένος, αλλά σύν με το ότι μία ακτή δεν είναι όμοια με τις υπόλοιπες. Μία δημόσια ακτή έχει διαφορετική αξία με μία άλλη παράκτια περιοχή η οποία βρίσκεται σε μια κατοικημένη περιοχή σαν παράδειγμα και θα έχει μεγαλύτερη αξία ενώ σε μια άλλη δημόσια περιοχή για να φτάσει κανείς πρέπει να κάνει χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων και θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Εφόσον πρόκειται λοιπόν για δημόσια κτήματα δεν θα πρέπει να δίδεται σε ορισμένους η εκμετάλλευση της περιοχής με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε κάποιον άλλον για μια διαφορετική περιοχή. Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τα δεδομένα τα οποία μας μεταφέρει ο αναφέρον εν μέρη είναι σωστά. Έχω εδώ μια έκθεση της Διεθνής Οργάνωσης για την Προστασία της Πανίδας που λέει ότι στα ερωτήματα τα οποία θέτουμε για την διεύρυνση των εμπορικών εγκαταστάσεων Υπάρχουν κάποια στοιχεία αριθμητικά τα οποία δεν βρίσκουμε εμείς ότι είναι σωστά και όχι μόνο εμείς. Συνεπώς λοιπόν δεν ξέρω ακριβώς πόσες είναι αυτές οι περιοχές που ανήκουν σε ευρύτερα δημόσια κτήματα, δημόσιες κτήσεις, πάντως είναι σαφές ότι πρόκειται για περιορισμένους πόρους. Ταυτόχρονα Θυμίζω ότι οι περιφέρειες είναι υποχρεωμένες ένα τμήμα των εδαφών αυτών να τα αφήνουν σε ελεύθερες ακτές. Στην Λιγουρία το 40% των παράκτιων περιοχών πρέπει να μείνει ακάλυπτο, στην Απουλία το 60% πρέπει να παραμείνει ακάλυπτο. Ε, έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι πράγματι οι παράκτιες αυτές περιοχές είναι περιορισμένος πόρος και σε αυτό προστίθενται και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γύρω από το ισπανικό θέμα, το νόμο τον ισπανικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται το θέμα. Αυτό το οποίο συνέβη τον μήνα Απρίλιο του 2013, αν δεν κάνω λάθος, όταν υπήρξε η ανακοίνωση της κυρίας Επιτρόπου Ρέντινγκ, είχαμε περιοριστεί σε μια πρώτη αξιολόγηση μιας κατάστασης ιδιαιτέρως περίπλοκης και αυτή η παρέμβαση ε, είχε προηγηθεί μιας εξέτασης του θέματος επί τη βάση του κοινοτικού δικαίου. Η Ισπανία έχει ξεκινήσει από μια διαφορετική αφετηρία. Δηλαδή οι ε, εκτάσεις αυτές ήσαν ελεύθερες, επολύθησαν, υπήρχε μέχρι σε κάποια φάση μια άγρια εκμετάλλευση αυτή, παράνομη θα έλεγα, και η ισπανική κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να σταματήσει τις δραστηριότητες αυτών των αυθερέτων παρανόμων εγκαταστάσεων και τελικά αναγκαστήκαμε ε, να αποζημιώσουν αυτούς τους ιδιώτες οι οποίες ε, στην ουσία μετετράπησαν από ιδιωτικές περιοχές σε περιοχές δημοσίας κτήσης. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι απόλυτα συμβατή η ισπανική περίπτωση με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Έχουμε λάβει αρκετές καταγγελίες ε, γύρω από την ισχύ και την αποτελεσματικότητα του νόμου για τις ακτές. Υπάρχουν κριτικές και τις εξετάζουμε. Πρέπει να πω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει αυτό το ερωτηματολόγιο σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τις δημόσιες παραλίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάνουμε τώρα μια συγκριτική μελέτη της κατάστασης της σα στα διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή στάση συμβατή ε, σε όλες τις χώρες. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και έχει αναφερθεί πάρα πολύ συχνά στην Ιταλία και έχει δημοσιευθεί. Όταν μιλούμε για τις Ιταλικές ακτές, μιλούμε για 30.000 επιχειρήσεις. Οι περισσότερες μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι οποίες ε, έχουν κάνει μια συμφωνία με τις Ιταλικές αρχές Γιατί προηγουμένως οι ακτές, οι παραλίε ήταν απολύτω ελεύθερες από τη διαχείριση, αν θέλετε, ή την οικονομική εκμετάλλευση. Οι επιχειρήσει αυτές με το Ιταλικό κράτος έχουν επενδύσει και έχουν ε, δημιουργήσει ένα τομέα ε, πραγματική ερωτική αριστεία. Από τη στιγμή που ο τομέας αυτός δεν αναπτύχθηκε σε καμία άλλη χώρα κατά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε στην Ιταλία. Θεωρώ ότι πρόκειται λοιπόν για ένα, μια επιτυχία made in Italy, λέει ο μιλητής. Διότι ο τρόπος αυτός δεν ακολουθήθηκε σε άλλες χώρες. Επομένως, σχετικά με την μετακίνηση των υπηρεσιών στην Ευρώπη, διαρωτώ με ποιον τρόπο μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στι παράκτητε περιοχέ, ε, θα μπορούσε να πάει να επενδύσει στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη χώρα, ιδιαίτερα του Βορρά. Ενώ αντιθέτω, μια γερμανική επιχείρηση μπορεί ωραιότατα να έρθει στην Ιταλία και να λάβει μια τέτοια παραχώρηση. Δεν υπάρχει λοιπόν αμοιβιότητα ή τουλάχιστον αμοιβιότητα που να έχει νόημα ε, προς την εφαρμογή δηλαδή της οδηγίας των υπηρεσιών. Τώρα, πάνω απ' όλα στο πλαίσιο της κρίσης και σε αυτήν τη λογική υπέβαλα και την αναφορά, θα πρέπει κανείς να δει την οικονομική κρίση. Μιλούμε για μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονη δυσκολία. Και δεδομένης της περιπλοκότητας του όλου προβλήματος, νομίζω ότι θα έπρεπε να το δει κανείς ε, πληρέστερα. Εγώ θα επιθυμούσα αυτές οι παραχωρήσεις ε, να διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο και απολύτως ευόμενη την επικουρικότητα, διότι οι ευρωπαϊκές αγορές διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και διακινδυνεύουμε ε, σοβαρές ζημιές και αρνητικό αντίκτυπο. Μιλούμε για τις παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο σε, άλλες, σε άλλους τομείς ε, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ε, οι Γερμανοί φίλοι μας ε, ήταν, απέκλεισαν τα δικά τους χωρικά ύδατα από τις παραχωρήσεις, ενώ εμείς ε, διαμαρτυρόμεθα μονίμως γιατί υπάρχει αυτή η πολύ διαφορετική μεταχείριση μεταξύ του Νότου, ημών, εν πάση περιπτώσει, και του φορά της Ευρώπης. Δεν θα ήθελα λοιπόν να θεωρηθεί η Ιταλία β' κατηγορίας, ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές ε, στο παρελθόν. Και, και στις περισσότερες περιπτώσεις ε, ο κίνδυνος περιορίζεται πάντα σε συγκεκριμένες χώρες. Και αυτό, αυτή η περιοριστική ερμηνεία δεν είναι καθόλου σαφής πάντως σε σχέση με τις περιοχές αυτές τα δύο τρίτα των ε, παρακτήρων περιοχών είναι, εξακολουθούν να είναι ελεύθερες. Νομίζω ότι κανείς θα έπρεπε να προσπαθήσει να βρει ένα σύστημα προστασίας αυτών των επιχειρήσεων. Ενδεχομένως μόνο για τις νέες παραχωρήσεις. Καθότι υπάρχουν παραλίες, καθότι οι δήμοι προχωρούν σε νέες παραχωρήσεις, εν πάση περιπτώσει αυτοί που ήδη είναι δικαιούχοι, να μπορέσουν τουλάχιστον να αποσέσουν την επένδυσή τους. Γιατί αυτές οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ε, στις οποίες αναφερόμουν έχουν αναλάβει σημαντικό βάρος δανείων ε, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν και στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που τους ε, χρειάζονται για να προχωρήσουν στη δραστηριότητά τους. Και μιλούμε για δάνεια 10-15 χρόνων ώστε να επικαιροποιήσει κανείς, να ανακαινήσει τις εγκαταστάσεις, τις πισίνες, το ό,τι είναι. Χρειάζονται λοιπόν, χρειάζεται χρόνος προκειμένου αυτές οι παραχωρήσεις να επανέλθουν και να εμπέσουν τελικά στην προσπάθεια και την επένδυση που έχει γίνει. Επομένως, δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης και της κρίσης και δεδομένης και της ιδιαιτερότητας της Ιταλικής, θα σας ζητούσα να το σκεφτούμε το ζήτημα σοβαρά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την απάντηση της Επιτροπής. Είναι σε δύο τμήματα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επιμείνω στο δεύτερο τμήμα της απαντήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί φαίνεται να μας προσφέρει κάποιες λύσεις για το πρόβλημα, διότι μας λέει ότι ε, το πρόβλημα των ε, επιχειρηματιών, των παραχωρησιούχων, σε περίπτωση παραχωρήσεων που ανανεώνονται αυτομάτως ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον βέβαια και οικονομικά είναι, ε, έχουν ληφθεί υπόψη τα συμφέροντα των ε, εμπλεκομένων, τα οικονομικά δηλαδή συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι βλέπω δηλαδή εδώ πέρα, μας λέει ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει ε, επαφές με τις ε, Ιταλικές αρχές σε αναζήτηση λύσης για το πρόβλημα. Αυτό που βλέπω δηλαδή στο πρώτο τμήμα είναι ότι μας εξηγεί η Επιτροπή την, ε, το νομικό πλαίσιο σε σχέση και με την οδηγία για τις παραχωρήσεις. Στο δεύτερο όμως τμήμα αναγνωρίζει και ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή μας λέει η Επιτροπή να αυτό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι το επιθυμητό. Γιατί δεν θέλουμε να κλείσουμε καμιά οικογενειακή επιχείρηση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θέλουμε να προξενήσουμε ζημιά οικονομική σε καμιά ευρωπαϊκή οικογενειακή επιχείρηση. Και έτσι προτείνουμε μία λύση. Αυτό μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ λοιπόν προτείνω σε εκ τούτου να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και παρακαλώ την, ε, τον πρόεδρο της Επιτροπής ή εμάς όλους αν χρειάζεται να απευθύνουμε μια επιστολή να ζητήσουμε, πάση περιπτώσει, κατεπηγόντως ε, με την Ιταλία, άλλωστε και η Επιτροπή ίδια το προτείνει, να ξεκινήσουν επαφές με την Ιταλία, να απευθύνουμε λοιπόν έκκληση για μια ταχύτατη ανάληψη επαφών και συνομιλιών με τις Ιταλικές Αρχές προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα. Άλλωστε, Βλέπουμε ότι υπάρχουν από ό,τι φαίνεται ανάλογα με την ανομή τάξη, κάποιες ε, ειδικές διατάξεις, ε, δυνατότητες για λύση στην Ευρώπη. Η θητεία μας βέβαια λίγη, το ξέρουμε αυτό, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον μέχρι τελευταία μας συνεδρίαση να λάβουμε και μια απάντηση, ενημέρωση για το αν έχουν ξεκινήσει αυτές οι συνομιλίες. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για οικογένειες που έχουν πάρει δάνεια και που ε, κινδυνεύουν να χάσουν τις παραχωρήσεις ενώ έχουν χρεωθεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει στην τελευταία μας στο συνεδρία να ενημερωθούμε αν έχουν ξεκινήσει έστω οι συνομιλίες. Παραμένει όπως λέω, όπως συστήνω, ανοιχτή η αναφορά και καλώ την Επιτροπή και την Ιταλία να αναλάβουν συνομιλίες για την εξέβρεση λύσεως, όπως θα μας προτείνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί διαβάζοντας το νόημα τουλάχιστον της έκθεσης της Επιτροπής, βλέπω, εάν το διαβάζω σωστά το νόημα αυτό, ε, ότι και η Επιτροπή αυτό ζητάει, να, γίνει, να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μπαλντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απευθύνω ένα χαιρετισμό και στον αναφέροντα που θίγει σημαντικό ζήτημα. Γιατί αφορά και σε παραλίες όχι μόνο Ιταλικές αλλά και όλες τη Μεσογείου. Το κατά πόσον είναι περιορισμένοι αυτή η φυσική πόροι ή σπάνιοι είναι αν θέλετε περισσότερο γλωσσικό ζήτημα και όχι ουσιαστικό. Προφανώς δεν υπάρχουν αναρρύθμιτες παραλίες αλλά δεν έχουν και όλες οι παραλίες την ίδια αξία. Εγώ είμαι από την Ίστρια όπου όλο και πιο λίγες παραλίες είναι ελεύθερες. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί η χρήση και η διαχείριση αλλά και να διατηρηθεί η κρατική, η δημόσια ιδιοκτησία, όπως και να διατηρηθούν ελεύθερες παραλίες. Ακούσαμε το μέγεθος αυτό του 70% των ελεύθερων παραλίων στην Πούλια, αλλά γιατί είναι έτσι, γιατί έτσι το επιθυμούν. Θέλουν ε, να έχουν ελεύθερες παραλίες και τους συγχαίρω τους κατοίκους της Πούλια και τις αρχές της. Τώρα η σύγκριση με την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κροατία ε, και εκεί υπάρχει το φαινόμενο. Και σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να χαιρετήσω τους φοιτητές της Τσέρα που μου θυμίζουν κάποιες ε, σπουδές, τις σπουδές μου. σχετικά με τους Ατσερεντίνοι οι οποίοι ίδρυσαν πολλές απικίες ε, στα εδάφη από τα οποία προέρχομαι εγώ και προχώρησαν σε μεγάλα έργα στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές και μιλούμε για ιστορία 2.000 ετών. Έργα λοιπόν σπουδαία και απικίες σπουδαίες που οι οποίες μας προσέφεραν θαλάσσιες και παραθαλάσσιες δουλειές σπουδαίες. Ήθελα απλώς να αναφέρω και αυτό, μια και είναι οι σπουδαστές εδώ παρόντες. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαλτίνη, λέει η Πρόεδρος. Δεν έχουμε... Α, ο κύριος Μοργάτη θέλει κάτι να απαντήσει. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, να συμπληρώσω απλώς. Θυμίζοντας ότι πρόσφατα το Ιδωλικό Κοινοβούλιο ψήφισε μια τροπολογία εξαίρεσης για την οδηγία υπηρεσιών για να κερδίσει λίγο χρόνο ακριβώς προκειμένου να επιλύσει αυτό το ευαίσθητο πρόβλημα. Η Κομισιόν τι θεωρεί για την τροπολογία αυτή και τη γνωρίζει επίσης την Κομισιόν γιατί αυτό δεν το κατενόησε από την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Επιτροπής. Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κι εγώ μία σκέψη που θα την υπέβαλα στην Επιτροπή. Μιλούμε για την γραπτή απάντηση της Κομισιόν σχετικά με τη διάκριση μεταξύ παραχώρησης του αγαθού, του ακινήτου και της υπηρεσίας. Εδώ μιλούμε λοιπόν για την παραχώρηση της υπηρεσίας τονίζει η Κομισιόν και όχι τόσο του ακινήτου περιουσιακού στοιχείου. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως αυτό το ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου, του κράτους, παραχωρείται υπό προϋποθέσεις και όρους που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένους περιοριστικές διατάξεις όπως αυτές στις οποίες αναφέρεται η Κομισιόν στην απάντησή της σχετικά με την τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τη διαχείριση του στοιχείου του περιουσιακού. Οι σημερινές παραχωρήσεις θαλασσίων χώρων υπάγονται σε κάποια σε κάποιες διαδικασίες και ιεραρχίες επαγγελματική δεξιότητα, κατάρτιση, εξειδίκευση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια για παράδειγμα της περιοχής. Υπάρχει μια ε, παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας αν θέλετε ελέγχου και, και καθαρισμού της παραλίας σεβόμενοι τις διατάξεις, ε, τις περιβαλλοντικές ε, που αφορούν ε, το θαλάσσιο χώρο και τον παράκτιο χώρο. Διατάξεις που αφορούν και στην πρόσβαση προς την θάλασσα. Διότι πέραν των ελεύθερων παραλιών έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή νομοθεσία στην Ιταλία που ακόμα και σε περίπτωση παραχωρήσεων προβλέπει την ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγαλό, στην ακτογραμμή. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι διατάξεις προς τις οποίες πρέπει να συμπορφώνεται η εκμετάλλευση και η παραχώρηση. Και όλα αυτά δεν είναι, δεν είναι τόσο αυστηρά συνδεδεμένα μόνο με την παραχώρηση της υπηρεσίας, αλλά με την διαχείριση ενός περιουσιακού στοιχείου όπως σας είπα. Επομένως είμαστε σε πεδίο λίγο διαφορετικό από το πεδίο στο οποίο υποτίθεται πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία υπηρεσιών. Και τέλος, σχετικά με την σπανιότητα των πόρων, δεν νομίζω ότι ο αναφέρον λέγει ότι είναι ενιολογικό ή γλωσσικό το πρόβλημα μεταξύ των πόρων, των σπανίων ή των απεριορίστων κτλ. Απλώς λέει ότι είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς ότι είναι περιορισμένη αυτή η πόρη. Όλοι οι πόροι, εν περιπτώσει, του πλανήτη είναι περιορισμένοι υπό κάποια έννοια. Σε σχέση όμως με έννοιες που μπορούμε να εξετάσουμε και να αναλύσουμε, πεπερασμένες σε περιπτώσει, οι παραλίες, τουλάχιστον οι δικές μας, είναι ένα στοιχείο της ε, περιουσίας της εθνικής μας με συγκεκριμένο μέγεθος και αριθμό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν η Κομισιόν τι προσέγγιση έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμή προκειμένου να εξακολουθήσουν αυτές οι επαφές και συζητήσεις μεταξύ της Ιταλικής κυβέρνησης και της Κομισιόν. Παρακαλώ. Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για τον πιθανό διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κρατομέλος ή στα κράτη-μέλη, φυσικά και είμαστε υπέρ. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από τον Επίτροπο Μπαρνιέ, απεδείχθη από τον Επίτροπο Μπαρνιέ σε μια συνάντηση στην οποία ήταν παρόν και ο Ευρωβουλευτής Μοργκάντη έτσι ώστε να υπάρξει μια, έγινε μια συζήτηση για να υπάρξει μια λύση. Συνειδητοποιούμε τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν και έρχομαι στο θέμα του προγράμματος για το 2020. Η οδηγία για τις υπηρεσίες έπρεπε να εφαρμοστεί στις 28 Δεκεμβρίου του 2009. Έπρεπε τότε να ξεκινήσουν δηλαδή οι διαδικασίες για την με ανταγωνιστικό τρόπο εκχώρηση αυτών των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης. Μετά πήγαμε στο 12, μετά στο 15 και τώρα πάμε στο 20. Και αν δεν είχε ε, ήδη παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω ακριβώς των προβλημάτων που υπάρχουν στην Ιταλία σε αυτό το επίπεδο, θα είχαμε καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να ξεπεράσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε το θέμα σαν παράδειγμα της διάρκειας των παρεχωρήσεων αυτών για εκμετάλλευση. Το άρθρο που ψηφίστηκε το 12 είναι το, πιο, ε, το λιγότερο επεξηγηματικό αν θέλετε, είναι κάτι που ε, πρέπει να εξαρτάται από το ύψος των επενδύσεων, πρέπει να είναι επαρκής η διάρκεια για να επιτρέψει την απόσβεση της επένδυσης. <clears throat> το πρόβλημα λοιπόν που έχει σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ξεκινήσει εν περιπτώσει αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών. Το θέμα δεν είναι μόνο η διάρκεια των παραχωρήσεων. Επί του θέματος της διάρκειας των παραχωρήσεων, όπως ήδη σας είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευέλικτη απαιτείται έλογη διάρκεια ανάλογα με το ύψος των επενδύσεων. Από το 9 μέχρι το 20 πάντως 11 χρόνια χωρίς ρυθμίσεις παραβιάζοντας ουσιαστικά την ισχύ της οδηγίας για τις υπηρεσίε είναι απαράδεκτο. Το συνειδητοποιούμε αυτό και αναζητούμε μία κάποια λύση και να ερμηνεύσουμε ε, όσο μπορούμε με ευρύτερο τρόπο με διασταλτικό τρόπο την οδηγία για τις υπηρεσίες αναλύοντας όπως σας είπα την κατάσταση στα κράτη-μέλη, συγκρίνοντας την κατάσταση και με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα καταλήξουμε σε μια ομοιογενή θα έλεγα γραμμή για όλα τα κράτη. Σχετικά τώρα για την παραχώρηση αγαθών και υπηρεσιών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι Πράγματι η βασική παραχώρηση είναι η παραχώρηση του συγκεκριμένου αγαθού, της έκτασης και λοιπά Αλλά καλύπτει και το θέμα των υπηρεσιών. Αν εδώ εφαρμόζεται άμεσα η οδηγία για τις υπηρεσίες και αν διευκρινίζονται μέσω της οδηγίας αυτής οι ρυθμίσεις για την εκμετάλλευση μιας υπηρεσίας και την παροχή μιας υπηρεσίας τόσο το καλύτερο σχετικά με τον περιορισμό των πόρων ή καλύτερα με τους λεγόμενους περιορισμένους πόρους. Κοιτάξτε, εμείς δεν νομίζω ότι ο όρος ε, περιορισμένη πόρη, δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπει πάρα πολλές ερμηνείες. Εμείς θεωρούμε ότι ε, οι παραλίες λόγω της φύσης τους είναι περιορισμένες. Πρόκειται δηλαδή για ένα αγαθό κρατικό, για ένα δημόσιο κτήμα. Ακριβώς λόγω του δημόσιου χαρακτήρα όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό για την εκμετάλλευση και την παραχώρηση. Ανεξαρτήτως από το θέμα του ύψους των οικονομικών πόρων θα επαναλάβω κάτι το οποίο έχει πει και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και το Συμβούλιο Υπουργών και η Ανώτατη Αρχή για τον Ανταγωνισμό. Πρόκειται για μια βασική αρχή την οποία θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας. Σχετικά λοιπόν με τους περιορισμένους πόρους, εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω, ότι κάθε περιφέρεια έχει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες να εκχωρήσει ένα ποσοστό των ελευθέρων παράκτιων περιοχών, 40%, 60% κτλ. Και θυμίζω ότι και κάθε παραλία έχει τη δική της αξία. Έχουμε πολλές καταγγελίες από πλευράς πολιτών που θα ήθελα να έχουν κάποιες παραχωρήσεις, όχι σε οδήποτε τυχαίο έδαφος του παράκτιου Ιταλικού εδάφους, αλλά σε συγκεκριμένες περιφέρειες γιατί κάποιο μέρος συγκεκριμένο έχει κάποια χαρακτηριστικά, έχει κάποιες ιδιότητες, έχει κάποια τοποθεσία ειδική. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση το δημόσιο κτήμα να παραχωρείται στον πρώτο τυχόντα. Ελπίζω να απάντησα στο θέμα που τέθηκε για τους περιορισμένους πόρους. Λοιπόν, ο αναφέρον ένα λεπτό αν θέλει κάτι να προσθέσει. Δεν είναι αλήθεια ότι στον πρώτο τυχόντα δίδονται παραχωρήσεις. Οι παραχωρήσεις ε, δίδονται με βάση κάποιους ε, επίσημους διαγωνισμούς, υπάρχουν αιτήσει οι οποίες κατατίθενται. Αφού γίνει λοιπόν ένας διαγωνισμός υπάρχουν συμμετοχές, δηλώσεις συμμετοχής και δίδονται κάποιες γέες προς παραχωρήσεις Πολλές φορές γίνονται πωλήσει των παραχωρήσεων αυτών από τον προηγούμενο στον οποίο είχαν παραχωρηθεί και ξαφνικά κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλές οικονομικές ζημίες. Απαιτείται να υπάρξει διάλογος. Συναντήσεις όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά με τους ίδιους αυτούς οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιες τέτοιες εκμεταλλεύσεις έτσι ώστε να εξηγηθεί στην κυβερνητική πλευρά το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για την Ισπανία τώρα. Παραδόξως αυτό το οποίο συνέβη στην Ισπανία το 88 όταν απαλωτριώθηκαν κάποιες ε, εκτάσεις από πλευράς ε, των ιδιωτικών συμφερόντων. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στην Ιταλία. Πολλές φορές ξέρετε ότι τα αυθαίρετα τα οποία έχουν χτιστεί, εγκαταστάσεις, δισκοτέκ, πισίνες, ε, γενικά διάφορες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αυστηρά ιδιωτικές. Και αυτό είναι προφανές. Αν πρέπει να επανέλθουν σε δημόσια χέρια αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προηγηθεί μία απαλωτρίωση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολλές δυσκολίες. Το να φανταστεί λοιπόν κανείς ότι ε, όλες οι παραχωρήσεις θα βγουν σε διαγωνισμό για παραχώρηση, για εκμετάλλευση ακριβώς, όλα αυτά μαζί γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανά περιοχή, ένα τοπικό περιβάλλον και υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στις αρχές και αυτούς που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση. Δεν μπορεί να αλλάξει βία το σύστημα. Ευχαριστούμε λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή. Η αναφορά από τις παρεμβάσεις ε, και τους ομιλητές που άκουσα όπως και από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ε, μας ανέφερε θέσεις που γνωρίζουμε, αλλά υπογράμμισε και το εκτιμώ, την ανοιχτή θέση που έχει η Κομισιόν απέναντι σε μια συμφωνία η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να προστατεύσει όχι μόνο τις περιοχές αυτές, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα. Η Κομισιόν προχωρά σε μια δραστηριότητα εξερεύνησης, αν θέλετε, ανείχνευσης σχετικά με τις περιοχές αυτές, ώστε να αποφευθούν ε, αποκλήσεις ε, ε, όπως αυτές που καταγγέλθηκαν δικαίου σημεί από τον αναφέροντα για, χώρες, για κρούσματα σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε ποιος τελικά θα είναι ο, ο ενιαίος και μη διακριτικός προσανατολισμός που θα υιοθετήσει η Κομισιόν απέναντι σε όλες τις χώρες, απέναντι σε τέτοιες de facto καταστάσεις. Εγώ είχα καθήκον να συνοψίσω λοιπόν τα όσα ακούστηκαν ώστε να τα ξαναυποβάλω προς την Επιτροπή για να λάβω κάποιες απαντήσεις πιο συγκεκριμένες ενδεχομένως πέραν δηλαδή του σύντομου γραπτού σημειώματος που λάβαμε. Να ευχαριστήσω όμως ε, τον αναφέροντα, την εκπρόσωπο της Κομισιόν και τώρα θα πάμε... Στο σημείο 6, αναφορά του Χαντριχ Χάλα, γερμανικής ηθαγένειας, που δεν είναι παρόν. Και δίνω το λόγο στον κύριο Ότινγκ της Επιτροπής Απασχόλησης. Σα ευχαριστώ. Στην υπόθεση αυτή έχουμε να κάνουμε με έναν Γερμανό, ο οποίος εργάζεται σε μια Ολλανδική εταιρεία ε, οικοδομική. Έχει το 2008 το Μάιο ένα ατύχημα με πόδι σπασμένο κτλ. Έχει καταρχάς μια πρώτη ε, αγωγή στι μετά στο Μαγδεμβούργο με επιβάρυνση της Ολλανδικής του ασφάλειας και από το 2011 έχει ε, σύνταξη αναπηρίας γιατί δεν μπόρεσε να ε, αποκατασταθεί πλήρως με την αγωγή το πόδι του. Εν τω μεταξύ από τον Μάιο του 2011 έχουν πέσει οι ε, παροχές έχει υπαχθεί στη, στο γερμανικό ασφαλιστικό σύστημα, είναι στο ελάχιστο των παροχών, έχει απευθυνθεί ανεπιτυχώς στο Γερμανικό Υπουργείο Εργασίας και τις άλλες αρχές. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βλέπουμε καμιά δυνατότητα για παρέμβαση, διότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν βλέπουμε να έχει παραβιαστεί εν προκειμένου. Το ζήτημα του κατά πόσον ένα ατύχημα καταχωρίζεται ως επαγγελματικό ατύχημα, επαγγελματική ασθένεια ή όχι, ανήκει καταρμοδιόταν στο κράτος μέλος και ως εν προκειμένου το Ολλανδικό κράτος. Ευχαριστώ κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ για την απάντηση την Επιτροπή. Θα πρέπει να δούμε λίγο και το πρόβλημα του αναφερομένου ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει από τον Άννα στον Καϊάφα στις γερμανικές αρχές απάντηση για το ποιος είναι αρμόδιος. Επομένως, εφόσον μας λέει, ότι η Ευρωπαϊκή, μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αρμόδια το Ολλανδικό κράτος, εάν θέλει να αναλάβει κάποια δράση δικαστικού τύπου να χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσο αναφερόμενος, θα πρέπει να στραφεί στις αρμόδιες αρχές του Ολλανδικού κράτους, να στήσει τη βοήθεια δικηγόρων και να διεκδικεί στα δικαιώματά του. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Ήταν σαφής η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να τον ενημερώσουμε. Τώρα αναφερόμενο ε, ότι έχει τις δυνατότητες αυτές να ζητήσει υποστήριξη από δικηγόρους κτλ. Το πρόβλημα στην αρχή φαινόταν αρκετά απλό, εφόσον με το εργατικό αυτό ατύχημα ε, έλαβε, την κατα... έλαβε την αγωγή στις κατοχώρες, θεραπευτική αγωγή κτλ. Και μετά φαίνεται ότι από ένα σημείο και μετά χάνει ο αναφερόμενος την επικοινωνία δεν μπορεί να βρει ποια είναι η αρχή αρμόδια με την οποία πρέπει να επικοινωνήσει και γι' αυτό νομίζω αν του υποδείξουμε ότι αρμόδιο είναι το, το κράτος των κάτω χωρών θα τον βοηθήσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος λέει πρόεδρος. Όπως προτείνει λοιπόν ο κύριος Γιάρ μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά αφού η Επιτροπή έδωσε απάντηση στον αναφερόμενο. Συμφωνούμε. Καλώς κλείνει αυτή η αναφορά. Και περνούμε στο σημείο 8. Danny Byrne. Παρόν. Και του δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Το ιστορικό της αναφοράς μου είναι τραγικό. Ε, έχει να κάνει με τον θάνατο του πατέρα του αδελφού μου και τριών ακόμη συγγενών το 1981 στα νυχτά του Ντονεγκάλ στην Ιρλανδία. Ένα ατύχημα όπου μια βάρκα μέσα στη νύχτα προσέκουσε πάνω σε βράχια. Έχασα, όπως είπα, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου και τρία μέλη του πληρώματος, διορθώνει η μου. Η αναφορά λοιπόν σε στόχο έχει, σαν αντικείμενο έχει το εξή. Όταν ε, βούλιαξε αυτή η βάρκα άφησε αναξιοποιητό και το τονάζ το αλλιευτικό που είχε προβλεφθεί. Ωστόσο, το 2001 ξεκίνησε ένα σύστημα, ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται ε, «Αβαρία στη θάλασσα» και επέτρεπε σε όποιον έχει χάσει ε, σκάφος στη θάλασσα να ανακτήσει την αντίστοιχη αλλιευτική άδεια. Εμείς με μεγάλη καθυστέρηση ενημερωθήκαμε, δεν λάβαμε επίσημη ενημέρωση παρότι ήταν η το μεγαλύτερο αλλιευτικό σκάφος αυτό του πατέρα μου που βούλιαξε το μεγαλύτερο αλληλευτικό της ε, Ιρλανδίας, ενώ άλλοι που είχαν τις κατάλληλες πολιτικές συνδέσεις ενημερώθηκαν προσωπικώς για την δυνατότητα αυτή ανάκτησης της άδεια. Και μάλιστα κάποιοι από τους δικαιούχους είχαν προκαταβολικά ενημερωθεί πριν ληφθεί η απόφαση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πρόβλημα στην ελευθερία της ενημέρωσης. Η οικογένειά μου και ο φαινόμενος καταθέσαμε διαμαρτυρία έγγραφη στη γραφείο του διαμεσολαβητή της Ιρλανδίας που επί τρία χρόνια διερεύνησε την υπόθεση. και διαπίστωσε ότι δεν είχε χειριστεί σωστά την υπόθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο Υπουργός την εποχή εκείνη και το προσωπικό του και άρα έδωσε δίκαιο στην οικογένειά μου. Η κυβέρνηση όμως απέρριψε την έκθεση του διαμεσολαβητή την εποχή εκείνη. Είναι η μόνη απόφαση διαμεσολαβητή που έχει απορριφθεί από κυβέρνηση στην Ιρλανδία. Και κατόπιν αυτού έγιναν συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο συζητήσεις πάρα πολύ εντατικές που ε, ακολουθούσαν περισσότερο κομματικές γραμμές και έτσι παραγνωρίστηκε η έκθεση του διαμεσολαβητή. Αυτό είναι και ο λόγος που με φέρνει μπροστά σας σήμερα. Έχουμε εδώ και τρία χρόνια μια νέα κυβέρνηση στην Ιρλανδία, η οποία όμως ε, δεν θεώρησε σκόπιμο να εφαρμόσει αυτή την έκθεση. Έχουμε κάποιους πρώην υπουργού που τώρα ανήκουν στην αντιπολίτευση και θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια από το κόμμα των εργατικών ενός υπουργού πριν από λίγα χρόνια που έλεγε ότι είναι απίστευτο ένα τέτοιο θέμα να φτάνει να περάσει τόσα χρόνια χωρίς να αντιμετωπιστεί είναι απαράδεκτο για την πολιτική μας ζωή και θα πρέπει ε, να παραδεχθούν οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης τα λάθη τους στη μη υλοποίηση της έκθεσης του διαμεσολαβητή. Επίσης από το Φίνα Γκέιλ, ένας ε, υφυπουργός ε, στην Μικτή Επιτροπή για την Αλία το 2010 δηλώνει «Δεν αντιλαμβάνομαι τι είναι αυτό που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση και το οποίο μας απαγορεύει, μας εμποδίζει από το να δεχθούμε τη συστάση του διαμεσολαβητή. Ο ε, η Εμρή O'Reilly που τώρα είναι η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής ε, έχει αναλάβει το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αποτίσω φορό τιμής όπως επίσης και στον Ευρωβουλευτή που έχει προωθήσει την αναφορά. Πάντως βλέπω ότι η κυβέρνηση Ιρλανδίας δεν θεώρησε σκόπιμο να απαντήσει πάνω απ' όλα να ανταποκριθεί στην έκθεση του διαμεσολαβητή και να την εφαρμόσει. Η Άννα Εμπραχάμ, αντίστοιχα διαμεσολαβητή στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει σημειώσει ότι τα πράγματα αυτά παραμένουν, τα ευρήματα αυτά παραμένουν ε, ανεφάρμοστα και από τότε που η Έμιρο Ράιλι ανέλαβε καθήκοντα Ευρωπαϊκή Ευρωπαίου διαμεσολαβητή ε, δεν έχει, αντικατασταθεί, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτή η έκθεση. Κύριε Χίκινς, ένα λεπτό για να απαντήσει πρώτα η Επιτροπή. Κύριο Σούτισερ. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπέρν για τις εξηγήσεις σας, για την αναφορά σας, τη μελετήσαμε προσεκτικά. Είδαμε και την έκθεση του Ιρλανδού διαμεσολαβητή όπως βλέπετε και από τη γραπτή μας απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάση κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους της Ιρλανδίας και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι κάτι το οποίο αφορά την ικανότητα του στόλου και των αλλιευτικών σκαφών στην Ιρλανδική θάλασσα. Το 97 το Συμβούλιο υιοθέτησε μία απόφαση για την αναδιάφρωση του, του αλλιευτικού τομέα και την εξισορρόπηση των αλλιευτικών ικανοτήτων. Δημιουργήθηκε ένα μόνιμο καθεστώς ελέγχου ανανέωσης των σκαφών. Η Ιρλανδία υπέβαλε ένα πολιετές πρόγραμμα για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει και το Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα αυτό το 1998. Στη συνέχεια, όπως και το απαιτεί η απόφαση, ενημέρωσε η Ιρλανδία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύστημα εισόδου-εξόδου, αλλά δεν ενημέρωσε για το πρόγραμμα των απολειών των αλλιευτικών σκαφών όπως απαντήσαμε και στην ερώτηση του κυρίου Χίγκιν στο 2006. Ο τρόπος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανή ε, να διορθώσει τις αποφάσεις είναι τα άρθρα 12 και 58 της Συνθήκης για τη διαδικασία επιπαραβάση. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποίησε την, ε, το πρόγραμμα αυτό, ήταν πια πάρα πολύ αργά, δεν ίσχυε το πρόγραμμα, έχει, έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που σταμάτησε να λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό ήταν ε, ένα περιορισμένο πρόγραμμα συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και αφορούσε ένα μικρό αριθμό πολιτών. Μια διαδικασία επί παραβάση λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρείται ευκταία. Είναι σαφές βέβαια και από την έκθεση του Ιρλανδού διαμεσολαβητή ότι υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις στην οικογένεια ε, του αναφέροντος γιατί δεν ήταν γνώστες της διαδικασίας αυτής. Μια διαδικασία επιπαραβάση στρέφεται κατά του κράτους μέλους χωρίς άμεσες οικονομικές ε, συνέπειες ωφέλει καλύτερα για τον αναφέροντα. Ως εκ τούτου θεωρούμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μία δράση παραλήψης βάρος του κράτους μέλους ε, θα ήταν χρήσιμη. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ κύριο Χίγκινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που κρίνατε παραδεκτή την αναφορά αυτή. Σχετικά με το σκάφος που ήταν η ιδιοκτησία της οικογένειας Μπάιν. Στις 31 Οκτωβρίου μετά το ατύχημα αυτό έμεινε με τα μικρά παιδιά ο κύριος Μπέρν Το επεισόδιο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Irish Skipper και στο Marine Times. Επίσης εξειδικευμένο έντυπο για τα θαλάσσια ζητήματα. Αλλά σε ό,τι αφορούσε την οικογένεια το επεισόδιο αφορούσε μόνο, ενδιαφέρονταν μόνο μάλλον δηλαδή για το επεισόδιο για να συνεχίσουν τη ζωή τους και τίποτε άλλο. Η οικογένεια Μπάρν δεν γνώριζε για πάρα πολλά χρόνια την ύπαρξη του συστήματος αυτού του Lost Όταν κινήθηκαν είχε πια σταματήσει το σύστημα. Μετά την άρνηση του Υπουργείου υπέβαλα στην κυρία Ρέιλι το ζήτημα στο διαμεσολαβητή η οποία πρότεινε 245.000 ε, ευρώ ε, αποζημίωση για την οικογένεια Μπάριν. Η τότε κυβέρνηση το απέρριψε αυτό το αίτημα και τα επόμενα αιτήματα. Η έκθεση του διαμεσολαβητή είναι τεράστιο έγγραφο, λεπτομερέστατο, σαφέστατο και δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, πρόεδρε, αλλά ένα βασικό έβριμα λέει είχαμε πολύ αρνητικές συνέπειες για την οικογένεια μετά την άρνηση για την υποβολή υπό το σύστημα αυτό, το οποίο είχε σχέση με την ε, σωστή ορθή διαχείριση. και το σύστημα δεν είχε δημοσιοποιηθεί επαρκώς το Lost at Sea. Επίσης υπήρχαν ρούντο ανεπαρκή αρχεία στα πλαίσια του συστήματος αυτού, το οποίο είναι θέμα της Ιρλανδικής ε, κυβέρνησης. Ο διαμεσολαβητής, ο Ιρλανδός, είναι θεσμός από την αρχή του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, δεν είδα ποτέ έκθεσή του, αίτημά του, γνωμοδότησή του να απορρίπτεται. Και εδώ έχουμε μια έκθεση που συνιστά ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο απόρριψης, ε, ε, εισήγησης του διαμεσολαβητή. Ε, έχουμε να κάνουμε με μια χείρα που έχασε τον άντρα της και αναγκάστηκε να μεγαλώσει μόνη της τα παιδιά της, το πόρισμα του διαμεσολαβητή είναι σαφές, θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ ο κύριος Γκάλαχρη, λέει η Πρόεδρος. Δεν επιθυμείτε το λόγο. Ο κύριος Higgins το περιέγραψε τέλεια, δεν θα να σας αφήσουμε περισσότερο χρόνο για ερωτήσεις. Ο κύριος Βαλέσνα, Σύντομη ερώτηση. Γιατί απέρριψε την έκθεση του διαμεσολαβητή η Ιρλανδική κυβέρνηση, με τι αιτιολόγηση. Ο λόγος, για να σας απαντήσω, είναι πολύ καλή ερώτηση σας. Ο λόγος ήταν ότι ενημερωθήκαμε για τους φακέλους δυνάμει της αρχής της σχετικής με την ενημέρωση ε, ενώ θα έπρεπε λοιπόν να μην έχει ξεκινήσει καν αυτό το σύστημα της ανάκτησης, ο Υπουργός ε, έκανε ε, το σχέδιο αυτό, αλλά παραχώρησε το 75% των αποζημιώσεων μόνο σε δύο, σε δύο δικούς του ψηφοφόρους. Και βέβαια ορίστηκε μια προθεσμία για την κατάθεση της αίτηση για τη συμμετοχή στο σχέδιο αυτό, πάρα πολύ σύντομη, και φοβήθηκαν ότι εάν δίναν στην κυρία Μπέρν τη χείρα τη δυνατότητα αυτή. Όλοι εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να ενταχθούν στο σχέδιο θα κατέθεταν τις αιτήσεις τους, θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας και έτσι θα έπρεπε να πληρώσουν πάρα πολλά λεφτά για αποζημίωση σε πολλούς άλλους που δεν τους υπολόγιζαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Ίσως Ίσως αν μπορεί να σας φανεί λίγο άσχετο, αλλά πάντως είναι απίθανη αυτή η ιστορία που βλέπουμε να μας εκτίθεται εδώ. Έχουμε να κάνουμε με ένα ε, κανόνα, μια οδηγία, μια διάταξη η οποία απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη αλλά δεν τους γνωστοποιείται. Και απλώς προτιμούνται ορισμένοι αποδέκτες. Ε, ρωτώ όμως πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον αναφερόμενο, γιατί αυτή είναι η ουσία και καλύτερα ποιο είναι εκείνο το επίπεδο ή το όριο το οποίο κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαραίτητο για να διαπιστώσει παραβίαση συνθήκων ή υποχρέωσης κράτους κτλ. Γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε λοιπόν έχουμε να κάνουμε προγράμματα υποστήριξη, χρηματοδότηση, επιδοτήσει, όποιο, όποιος κανόνας βγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατίθεται πρέπει να ε, αποτελεί αντικείμενο πληροφόρησης για τον πιθανό δικαιούχο. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τον αναφερόμενο ή ποιο είναι αυτό το όριο ε, το οποίο ενδεχομένως παραβιαζόμενο οδηγεί σε μια διαδικασία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πρόεδρος. Μπορεί η Επιτροπή να δώσει μια απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως δεν είναι ζήτημα ορίου, αλλά η διαδικασία ε, επί παραβάση θα ήταν μια διαδικασία κατάλληλη για την αντιμετώπιση κράτους μέλους το οποίο παραβιάζει ευρωπαϊκό δίκαιο. Εδώ δεν βλέπουμε να έχει θεσπιστεί ευρωπαϊκό δίκαιο με το εν προκείμενο σύστημα για την ανάπτυξη της άδεια, διότι δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα δεν υπάρχει, α, και εντωμεταξύ δεν υπάρχει πλέον αυτό το σύστημα και δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε πλέον στην Ιρλανδία την ε, παραβίαση, διότι δεν υφίσταται πλέον αυτό το σύστημα αποζημίωσης. Δεν ξέρω εάν δυνάμει του Ιρλανδικού νόμου έχει κάποια άλλη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια ο αναφερόμένο στα Ιρλανδικά δικαστήρια, αλλά το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν βλέπω να μπορεί να αξιοποιηθεί στην περίπτωση αυτή και πάντως όχι η διαδικασία επί Ο κύριος Σίκη. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και για τις ε, σωστές ερωτήσεις σας. Τι ακριβώς θέλουμε. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη για την χείρα που έχασε τα παιδιά της, τον άντρα της, τους συγγενείς της, την περιουσία της. Εμείς θέλουμε η Επιτροπή Αναφορών να στείλει μια επιστολή στην Ιρλανδική κυβέρνηση και τον Σάιμον Κόφιλντ, τον τέος Υπουργό Αλίας, και να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της γιατί μια σύσταση έλογη σε σχέση με αποζημίωση προς την χείρα 235.000 ευρώ αγνοήθηκε πλήρως και να ζητήσουμε από τις Ιρλανδικές αρχές να λάβει σοβαρά υπόψη τους, να λάβουν υπόψη τους ε, την εφαρμογή της πρότασης του Ιρλανδού Ομπούτσμαν. Εφόσον συμφωνείτε λοιπόν λέει η Πρόεδρος μπορούμε να υιοθετήσουμε την πρόταση την οποία έκανε ο κύριος Χίγκινς, να στείλουμε μια επιστολή δηλαδή στις Ιρλανδικές αρχές και να ζητήσουμε να αποκατασταθεί η συγκεκριμένη κατάσταση γιατί πρέπει να αναζητηθεί μία λύση. Συνεπώς λοιπόν η αναφορά παραμένει ανοιχτή και θα στείλουμε επιστολή προς τις Ιρλανδικές αρχές. Ευχαριστώ τον αναφέροντα για την παρουσία του. Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχε παραμείνει ανοιχτό ένα σημείο της ημερησίας διατάξεως ε, και αν θέλετε μπορούμε να το δούμε τώρα κάτι δεν δουλεύει κάποιο κανάλι της διερμηνίας δεν λειτουργούσε. Κύριε Βαλέσα, έλεγα πρόεδρε, μια και τώρα ολοκληρώσαμε με τις υποβολές ε, των αναφορών και πριν από την ανάλυση της μελέτης να μιλήσουμε για το θέμα της ε, άκτα αν θέλετε να το κάνουμε τώρα, αν θέλετε να το κάνουμε στο τέλος, όπως μου πείτε Πρόεδρε. I think we can now the item because... hey, ε, πρόεδρος, μπορούμε τώρα να το συζητήσουμε αυτό. Ελπίζω, λέει η πρόεδρος, ότι δεν θα είναι μακροσκελές. Όχι πρόεδρε, δύο-τρία λεπτά θα χρειαστούμε στο δεύτερο παράρτημα των πρακτικών αναφέρεται η τοποθέτηση της μειοψηφίας σχετικά με την αποστολή στην Γαλλικία. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, διότι έτσι είχε αποφασιστεί, αλλά αυτό που δεν συμφωνούμε στο Λαϊκό Κόμμα είναι να αναφέρεται και τα πρακτικά της 14 Ιουνίου διότι δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται αυτό το έγγραφο εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι η έκφραση της ε, τοποθέτησης της μειοψηφία. Ένα έγγραφο 12 σελίδων, το, επί του οποίου δεν είχαμε συμφωνήσει καμία περίπτωση για το παράρτημα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το παράρτημα αυτό από τα πρακτικά και να αναφέρεται μόνο η τοποθέτηση της μειοψηφίας. Θέλει κάποιος κάτι να σχολιάσει, λέει ο πρόεδρος. Ναι, έχει δίκιο, πρόεδρε. Έχει δίκιο. Yes, okay, he's right, uh, Ωραία, εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά την περασμένη φορά είχαμε αποφασίσει να τοποθετήσουμε στο παράρτημα την ε, άποψη της μειοψηφίας. Η οποία πρέπει να παραμείνει στο παράρτημα. Eh, eh, eh, Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον τίτλο, λέει η Πρόεδρος. Όχι διακόπτει ο μιλητής. Όχι, Πρόεδρε, δεν είναι ο τίτλος το πρόβλημα. Είναι η άποψη της μειοψηφία που εμφανίζεται και προς το οποίο εμείς δεν διαφωνούμε, γιατί έτσι είχαμε συμφωνήσει, αλλά υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας 14 Ιουνίου του 2014 λέει ο μιλητής 12 σελίδων που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την άποψη της μειοψηφία. Κανένα πρόβλημα και καμία διαφωνία για την άποψη της μειοψηφία, αλλά αυτό το έγγραφο εργασίας, Πρόεδρε. Yes, it was clear. We have to put among the... ε, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι θα συμπεριλαμβάναμε την ε, άποψη της μειοψηφίας στο παράρτημα. Συμφωνείτε? Όχι. Ε, πρόεδρε, δεν ξέρω αν καταλάβα καλά. Ο κύριος τουργάιθ και εγώ καταλάβαμε ότι μπορούμε την μειοψηφούσα άποψη να την συμπεριλάβουμε. Αλλά αυτό το έγγραφο εργασίας όχι. Δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά. Ωραία λέει πρόεδρος. Άμα είναι τώρα σαφές το πράγμα, ας πάμε. Καθότι εγκρίναμε τα πρακτικά με την τροπολογία αυτή το σημείο 2, άρα μπορούμε να πάμε στο σημείο 9. για την παρουσίαση της ε, μελέτης σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Η κυρία η κυρία Βαλεστέρος έχει το λόγο, παρακαλώ. to... Η οποία θα μας κάνει μια παρουσίαση PowerPoint. Um... Καλησπέρα σας. Η συνάδελφος ε, Μανουέλα Κανέτα και η υποφαινόμενη Βαλεστέρος εργαζόμαστε σε ένα γραφείο για παροχή νομικών συμβουλών, πολιτικών συμβουλών για θέματα του ευρωπαϊκού δικαίου, κυρίως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε, Έχουμε αναλάβει θέματα αναφορών, ε, περιβάλλοντος, θεμελιωδών ελευθεριών και έχουμε ιδιαίτερως έρθει για να σας μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Πού είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας κάλεσε να αξιολογήσουμε εάν η πρωτοβουλία των ε, πολιτών, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ε, συνιστά αποτελεσματικό μέσον συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας καλεί να εξετάσουμε το πώς λειτουργεί, εάν Αξίζει τον κόπο όλης αυτής της διαδικασίας για τον οργανωτή. Αν είναι επαρκώς δημοκρατική, αν είναι αρκετή η δημοκρατία, αν αρκεί το να ζητήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση ή αν ενδεχομένω χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία. Γιατί ερχόμαστε τώρα να σας μιλήσουμε. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει και επιβεβαιώσει πως θα δημοσιευθεί στις 20 Μαρτίου μια, Ευρωπαϊ... μια ανακοίνωσή της για τις ε, πρώτες επιτυχής ευρωπαϊκής και πρωτοβουλίες πολιτών. Γίνονται ακροάσεις δημόσιες από την επόμενη εβδομάδα και από την υποβολή της ανακοίνωση ε, μέσα σε τρεις μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει σε μια αξιολόγηση εάν θα οδηγηθούν, θα ε, προκύψουν από τις πρωτοβουλίες αυτές των πολιτών νομοθετήματα, προτάσεις νομοθετικές ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να προσφέρει επιχειρήματα τόσο νομικά όσο και πολιτικά, πολιτικές επιλογές. Δεν έχει υποχρέωση να αναλάβει δράση, να προτείνει νομοθέτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει όμως υποχρέωση να απαντήσει στους πολίτες να αιτιολογήσει. Ο άλλος λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι ότι μέσα σε ένα μήνα από την εκκίνηση του εγχειρήματο βρήκαμε κάποια, καταλήξαμε σε κάποια ενδιάμεσα συμπεράσματα τα οποία καταγράφουμε στην ενδιάμεση έκθεση και ήρθαμε να σας τα παρουσιάσουμε. Ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμα για τα περαιτέρω βήματα που σας παρουσιάσαμε και έτσι θα σας δώσουν μια επισκόπηση του πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. στο μέλλον πρωτοβουλίε των πολιτών που δεν στεφόνται με επιτυχία θα μπορούσαν να περνούν σε συζήτηση ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να τα συζητά τα θέματα αυτά και να τα αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένω με τη μορφή των αναφορών ή και με τη μορφή νομοθετικής ε, πρωτοβουλίας όπου θα ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση νομοθετική, να καταθέσει πρόταση δηλαδή ε, για μια πρωτοβουλία, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν έχει λάβει επαρκή υποστήριξη με υπογραφέ. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν του στόχους της μελέτης, τη μεθοδολογία μας και πάνω απ' όλα τα προκαταρκτικά μας ευρήματα. Ο στόχος της μελέτης ήταν η εξέταση των προσκομμάτων που αντιμετωπίζει ο διοργανωτής όταν ε, ετοιμάζει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Εξετάζουμε και πιθανές λύσεις και τις παρουσιάζουμε βέβαια και στην ενδιάμεση έκθεση και σε μεταγενέστερο σχέδιο θα καταθέσουμε και συγκεκριμένες συστάσεις για να βελτιωθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Το δουλειά μας την κάναμε ως εξής μεθοδολογία. Κοιτάξαμε όλο το υλικό που υπάρχει στην υπόθεση αυτή, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μελετήσαμε τις απόψεις που μας έδωσαν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Συζητήσαμε, προσεγγίσαμε πάνω από 17 διαφορετικούς οργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών που μας είπαν τι είδους προβλήματα αντιμετώπισαν, πώς τα βλέπουν, τι είδους λύσεις τα έβρισκαν. Συζητήσαμε με τις εθνικές αρχές για το ποιες χώρες ε, παρουσιάζουν ή τι είδους ε, προβλήματα βλέπουν ανάλογα με τη χώρα στις διάφορες φάσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Συζητήσαμε με εκπροσώπους διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωβουλευτές, γραμματεία της, γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε γραμματεία της Επιτροπής των Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σε μεταγενέστερο στάδιο μία ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μας ε, συνδράμει στην κατάρτιση των συστάσεων ειδικοί εν προκειμένου, νομομαθείς, αλλά και ειδικοί στην, σε θέματα πολιτικής, στη συμμετοχική δημοκρατία. Και τώρα η συνάδελφος θα παρουσιάσει το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον κομμάτι της έκθεσής μας που είναι η τα προκατακτικά ευρήματα. Ευχαριστώ πολύ η Μάρτα. Μέσα σε ένα μόλις μήνα καταφέραμε να καταγράψουμε πολλά θέματα από τα όσα μας είπαν οι εμπλεκόμενοι, ίσως και με πιο πολλές λεπτομέρειες να σας είναι πιο ενδιαφέροντα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στις φάσεις της οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Εκεί βρίσκονται τα πιο πολλά προβλήματα, αλλά και σε μεταγενέστερα στάδια, σε όλη τη διαδικασία και από τα χαρακτηρίζουμε εγκάρσια ζητήματα. Βλέπετε εδώ τον κατάλογό τους. Θα κοιτάξω τον, τα σημεία 2, 3, 5 και 7 σε περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ βλέπετε τα 8 σημεία, τα προβλήματα όπως έχω, τα έχουμε ομοδοποιήσει. Θα περάσω τώρα πιο γρήγορα στα υπόλοιπα σημεία και ιδιαίτερα το ζήτημα, δηλαδή τα προσκόμματα που βλέπουν στην πιθανή υλοποίηση αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών που μας επισημαίνουν ε, οι συνομιλητές μας είναι οι πιθανότητε για προσωπική ευθύνη. Εδώ έχουμε να κάνουμε τα σημεία 1 και 6, προσωπική ευθύνη αλλά και προστασία προσωπικών δεδομένων, γιατί δεν υπάρχει ε, ένα σύστημα συγκεκριμένο. Υπάρχουν ε, ένα, εξ, ένα έως έξι άτομα τα οποία μπορεί να είναι υπόλογα για οποιαδήποτε δραστηριότητα ε, που, που, αναλα, αναπτύσσουν μέσα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ιδιαίτερα ο πρόβλημα είναι αυτό της στήρησης της νομοθεσίας σχετικής με την προστασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν δύναμη βέβαια του εθνικού δικαίου. Πολλοί μας λένε ότι είναι πολύ κοπιαστικό να οργανωθούν και τα γραφεία ε, κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ο εξοπλισμός ασφαλείας, πυρασφάλειας και ούτω καθεξής που απαιτείται για την διακράτηση των, εγγράφων με τις υπογραφές. Επίσης έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση, με την πληροφόρηση και την υποστήριξη που υποχρεώνει η νομοθεσία στο κάθε, στο κάθε κράτος να προσφέρει ο διοργανωτής της πρωτοβουλίας, γιατί εκεί είναι πολύ περίπλοκες οι διατάξεις. Και μια τελευταία παρατήρηση σχετική με την άμεση η απευθείας δημοκρατία που σας ανέφερε και η Μάρθα στην πρώτη διαφάνεια, γιατί αν δηλαδή είναι αρκετή αυτή η συμμετοχική δημοκρατία, να αναπτύσσεται επαρκώς και αν χρειάζεται κάποια αλλαγή στο σύστημα της πρωτοβουλίας των πολιτών. Αυτά όλα ανάλογα και με τα όσα θα σας παρουσιάσουμε στα προκτακτικά ευρήματα, γιατί βέβαια ηρωπείται δυνάμει του άρθρου 11 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, μπορεί να οδηγήσουν σε ανάγκη για τροποποίηση. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σα αναφέρω τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτέ. Καταρχά, το θέμα τη θέσπιση, τη εκκίνηση μια πρωτοβουλία, πώ να βρουν δηλαδή κάποιον ε, ε, εταίρο στα κράτη-μέλη, αν ε, ένα θέμα του ενδιαφέρει, πώ μπορούν να αναπτύξουν τη δραστηριότητα τη πρωτοβουλία και σε άλλα κράτη-μέλη. Με ιδιαίτερα επενετικά λόγια αναφέρθηκαν στην, ε, στο ρόλο τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που προάγει τι ανταλλαγέ και τι επαφέ μεταξύ των διοργανωτών και αντίστοιχα δυνατότητε για την ανάπτυξη πλατφόρμα επικοινωνία ε, χάρη στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω αναφέρονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μπορούσε να του βοηθήσει να επικοινωνούν μεταξύ του από το ένα κράτο στο άλλο. Ένα άλλο ήταν η χρηματοδότηση. Είναι ένα πολύ δαπανηρό ε, μέσων αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών από ό,τι μας λένε. Μας λένε ότι μπορεί να κοστίσει έως και ένα εκατομμύριο ευρώ η οργάνωση ε, μιας επιτυχούς πρωτοβουλίας των πολιτών, δηλαδή ένα ευρώ η κάθε υπογραφή και αυτό σημαίνει ότι διστάζουν ε, οι διοργανωτές όταν βλέπουν πόσο μεγάλο κόστος συνεπιφέρει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και ιδιαίτερα διστάζουν όταν ε, διαπιστώσει κανείς πόσο διαφορετικές είναι οι συνθήκες για μια πρωτοβουλία πολιτών και μια πρωτοβουλία οργάνωσης. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθούν αρκετοί πολίτες να διαθέσουν τα σχετικά κονδύλια. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο θα μας απασχολήσει και στην παρουσίαση των τελικών συστάσεων, στην τελική φάση της ε, έκθεσης μας, ίσως θα μπορούσε να εξευρεθεί μια δυνατότητα χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό ή και εθνικό επίπεδο ή να εξευρεθεί ένα σύστημα για αποζημίωση των εξόδων, επιστροφή εξόδων. Ένα άλλο θέμα ίσως πιο γρήγορα ακόμα, η ενημέρωση και η υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει ορατότητα στους διοργανωτές. Μας λένε ότι ήταν πολύ χρήσιμη η υποστήριξη από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως χρειάζονται ακόμη περισσότερη ε, υποστήριξη, έχουν πολύ περισσότερες ανάγκες από αυτό που έλαβαν. Θεωρούν ότι δεν είναι επαγγελματίε των εκστρατιών και μια πρωτοβουλία, είναι ε, ούτως υπήν ε, κοινοί άνθρωποι, απλοί πολίτες και θα ήθελαν περισσότερη υποστήριξη και τεχνογνωσία. Η ορατότητα επίσης, η δημοσιότητα και η ορατότητα και τι σημαίνει αυτό. Μας λένε οι συνομιλητέ μας ότι όταν ξεκινούν για μια εκστρατεία χάνουν πολύ χρόνο και πόρους να εξηγήσουν πρώτα απ' όλα τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, τι είδου εργαλείο είναι αυτό, τι σημαίνει η συλλογή των ε, υπογραφών. Πρώτα εξηγούν αυτό και μετά ξεκινούν την εξήγηση του θέματος που τους ενδιαφέρει να αναπτύξουν, να αντιμετωπίσουν σε μια πρωτοβουλία πολιτών του συγκεκριμένου ζητήματος δηλαδή. Και άρα καλούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για αυτό το σύστημα, για αυτό το μέσο, πέραν των επιμέρους ζητημάτων. Και επίσης πολλοί μας ανέφεραν ότι η εκστρατεία που ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ευρωεκλογές θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς να πλησιάσει τους πολίτες και να τους ενημερώσει, να τους ευαισθητοποιήσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δικαιώματα. Και επίσης οι ακροάσεις που αναμένεται να γίνουν μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα στην ευόδοση επιτυχών πρωτοβουλειών πολιτών, γιατί είναι μια ευκαιρία για την ενίσχυση της πρωτοβουλίας, της πρωτοβουλίας των πολιτών ως μέσου και όχι της ε, κάθε μίας επιμέρους πρωτοβουλίας και θεματολογίας. Προχωρώ στην πρώτη φάση που εντοπίσαμε, που είναι η καταχώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα λοιπόν έχει ε, δυνάμει της, ε, του σχετικού άρθρου της συνθήκης και των κανονισμών την ε, προϋπόθεση της στήρης ορισμένων κριτηρίων, τα οποία πρέπει να αξιολογήσει και μετά να καταχωρήσει τη σχετική πρωτοβουλία εφόσον πληρεί τα κριτήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο μετά ξεκινάει η συλλογή των πληροφοριών. Από τις προϋποθέσεις λοιπόν για την καταχώρηση μιας πρωτοβουλίας πολιτών, ε, ένα από τα κριτήρια και είναι και αυτό το που παρουσιάζει πιο πολλές δυσκολίες έχει να κάνει με τη νομική βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η κάθε πρωτοβουλία πολιτών. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει για τις σχετικές αρμοδιότητες τους πολίτες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν μια πρωτοβουλία. Εδώ ακριβώ είναι το σημείο τριβή, γιατί δεν έχουν την κατάλληλη γνώση οι οργανωτές των πρωτοβουλειών και πιστεύουν ότι χρειάζεται και περισσότερη σαφήνεια ως προς τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, έχοντας ε, δει από τις εμπειρίες ε, που έχουν ήδη συλλέξει ε, οι διοργανωτές των πρωτοβουλειών πολιτών, αλλά και τις απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπουμε ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια στην δημοθεσία. Άλλωστε υπάρχει και εκρεμή υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που άπαξ και καταλήξει σε τιμιγορία μπορεί να μας δώσει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία θα σωματώσουμε στη τελική φάση της έρευνας. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, πάλι στην νομική βάση, είναι η εξέταση σε δύο στάδια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λέμε ότι πρόκειται για δύο στάδια. Στάδια, γιατί είπαμε ότι πρώτα πρέπει να γίνει καταχώρηση και μετά, όπως σας είπε νωρίτερα η Μάρτα, εφόσον θεωρηθεί παραδεκτή επιτυχής η πρωτοβουλία, συλλεγούν δηλαδή οι υπογραφές, τότε κατατίθεται αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με την, από πλευρά τη αποφασίζει αν θα δώσει συνέχεια, αν δηλαδή θα προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από επαληθεύσει που πρέπει να γίνουν στην αρχή και άλλα περίπλοκα ζητήματα που εμπλέκονται εδώ. Αλλά όσον αφορά την τωρινή μας παρουσίαση θα τα αφήσω κατά μέρους. Όμως την τελική μας ε, ανάλυση θα τα δείτε σε πιο πολλές λεπτομέρειες. Το θέμα της μετάφρασης έχει τεθεί επίσης. Ε, αυτό είναι κάτι που ε, αντιμετωπίσαμε σχετικά σύντομα. Υπάρχει καθήκον μετάφρασης του κειμένου και του κειμένου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ένα επιπλέον βάρος για αυτούς οι οποίοι συλλέγουν τις υπογραφές. Μετά από την καταγραφή λοιπόν οι οργανωτές έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα σύστημα συλλογής υπογραφών online. Έτσι λοιπόν θα συλλέξουν υπογραφές και αν αποφασίσουν να συλλέξουν τις διαδικασίες έτσι θα πρέπει να δημιουργήσουν το λεγόμενο OCS, Online Σύστημα Συλλογής Υπογραφών θα πρέπει να υπακούει το σύστημα αυτό σε συγκεκριμένες προδιαγραφές έτσι ώστε να είναι ασφαλές και αξιόπιστο. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει δυσκολίες, υπάρχουν και αρκετά εμπόδια, εμπόδια τεχνικής φύσεως, τα οποία δεν θα σταθώ στην παρούσα φάση. Πρέπει να πούμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να καλύψει τις ανάγκες αυτής της φάσης Ταυτόχρονα όμως η πιστοσύνη του συστήματος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει και σε μεμονωμένα κράτη-μέλη, γιατί ισχύουν στην παρούσα φάση διαφορετικοί κανόνες στα διάφορα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία για τους οργανωτές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι έτοιμο ε, το κείμενο, πρέπει να επιλέξουν ένα σύστημα συλλογής υπογραφών, πρέπει να πιστοποιηθεί από τα κράτη-μέλη και μπορούν να ξεκινήσουν να συλλέγουν τις υπογραφίες. Στα σημεία 1 και 4 απαιτούνται ακριβώς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις και εδώ υπάρχουν περαιτέρω εμπόδια. Το πρώτο εμπόδιο είναι η προθεσμία για την σύλλογη υπογραφών που σύμφωνα με τον κανονισμό είναι 12 μήνες. Κάποιοι πιστεύουν από τους οργανωτές τους πιθανούς ότι είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άλλη ο ελάχιστος αριθμός των υπογραφών ανακράτος μέλος. Απαιτείται ένα συγκεκριμένο ποσοστό έτσι ώστε να χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Έχουν τεθεί κάποια όρια λοιπόν σύμφωνα με τον κανονισμό στα παραρτήματα και ανταποκρίνονται σύμφωνα με συγκεκριμένες εξισώσεις τα ποσοστά των εδρών που έχει το κάθε κράτος στο κοινοβούλιο. Το σύστημα αυτό όμως δεν λειτουργεί ικανοποιητικά μέχρι τώρα. Διαφορετικοί αριθμοί υπογραφών απαιτούνται σε χώρες που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό και γι' αυτό ε, απαιτούνται διαφορετικά ποσοστά για τον αριθμό των 7 χωρών που είναι ο ελάχιστος αριθμός χωρών. Υπάρχουν και άλλα κάποια θέματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια στη συλλογή ε, ε, των υπογραφών που θα εξετάσουμε σε μία ιστερότερη φάση. Μπορούμε αν θέλετε να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το θέμα της συλλογής των υπογραφών και ιδιαίτερα με την διαδικασία της υπογραφής. Α, υπάρχουν διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις ε, για τη συλλογή των υπογραφών και την επιβεβαίωσή τους. Υπάρχουν χώρες που ζητούν στοιχεία ταυτότητας και χώρες που ζητούν άλλου είδους στοιχεία για τη συμμετοχή και υπογραφή αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών. Τέθηκαν αρκετές ανησυχίες από τους οργανωτές έτσι ώστε να ε, μην υπάρχει πρόβλημα για τις χώρες που απαιτούν στοιχεία ταυτότητας. Πολλοί πολίτες είναι πολύ διστακτικοί για να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Έτσι λοιπόν και ιδιαίτερα μετά από τα σκάνδαλα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών οι ε, πολίτες συνειδητοποιούν ακόμα ε, περισσότερο τα θέματα της προστασίας ε, της εμπιστευτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων. Υπάρχει έλλειψη λοιπόν εναρμονισμού στις διάφορες χώρες και αυτό σημαίνει για τους οργανωτές ότι θα πρέπει να υπάρξει αρκετή έρευνα έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις διάφορες απαιτήσει και να προετοιμαστούν με διαφορετικό τρόπο αναχώρα. Κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε είναι το θέμα των ταυτοτήτων και η απόσυρση συγκεκριμένα των ταυτοτήτων έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, απάτες όταν ε, συλλέγονται υπογραφές το θέμα είναι βασικά τα δεδομένα αυτά να συλλέγονται με σωστό τρόπο, εμπιστευτικά να μένουν και δεύτερον προσπαθούμε να καταλήξουμε αν είναι δυνατόν σε μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή, εναρμονισμένη ευρωπαϊκά, έτσι ώστε οι οργανωτές να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σύστημα λειτουργίας της συλλογής των υπογραφών. Κάποιοι εμπλεκόμενοι θεωρούν ότι ε, θα πρέπει να ε, γίνουν κάποιες διευκρινήσεις και για τους ε, εκπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων που θα ήθελαν να πάρουν μέρος στη συλλογή αυτή των υπογραφών. Τώρα για την απόδειξη κατοικίας. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και μιας και τα συστήματα όπως είπα δεν είναι συντονισμένα μεταξύ τους, κάποιοι ε, πολίτες δεν μπορούν ουσιαστικά ε, να πάρουν μέρος. Ιδιαίτερα Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε τρίτες χώρες. Αυτό φαίνεται τεχνικό σαν θέμα, αλλά δείχνει ότι δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα υπογραφής. Κλείνοντας, και μετά από τις δύο τελευταίες φάσεις το ένα θέμα είναι ο έλεγχος των διαδικασιών από πλευράς των κρατών μελών. Μετά από τους 12 μήνες οι οργανωτές στέλνουν τα αποτελέσματα στα κράτη-μέλη και το κράτος μέλος το συγκεκριμένο επαληθεύει τις υπογραφές και εκδίδει ένα πιστοποιητικό προς τους οργανωτές με τον ακριβή αριθμό των εγκεκριμένων ψήφων Εφόσον είναι λοιπόν στα επίπεδα που απαιτείται ε, η καταμέτρηση προωθείται. Αυτό συμβαίνει τώρα γιατί ξέρετε οι πρώτοι οργανωτές τέτοια συλλογή υπογραφών βρίσκονται στη φάση της επαλήθευσης και είδαμε ποια εμπόδια έχουν έρθει στην επιφάνεια και προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε ανάλογα με τη χώρα. Στην τελευταία φάση της μελέτης αυτής, όταν συμμετέχουν περισσότερα μέλη στη διαδικασία ελέγχου, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε και περισσότερα προβλήματα και εκκρεμότητες. Η τελική φάση που είναι το, η τελική μας διαφάνεια είναι η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αποτελέσματος της συλλογής των υπογραφών. Επιβεβαιούνται τα, οι τρεις φάσεις, τα τρία βήματα, ε, ξέρετε ότι πρακτικά ε, θα οργανωθεί η πρώτη ακρόαση. Θα δούμε τον επόμενο μήνα πώς θα καταλήξει η πρώτη αυτή πρωτοβουλία. Και στην τελική μας έκθεση το μήνα Μάιο θα έχουμε ελπίζω εντοπίσει και άλλα προκαταρτικά θέματα και εκκρεμότητες. Ε, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω στην παρούσα φάση, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, για την παρουσίασή σας και για την μελέτη. Ας ακούσουμε ίσως τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μαγιστέρος και την κυρία Κανέτα για την παρουσίαση αυτή. Εμείς ε, <clears throat> χαιρετίζουμε την μελέτη αυτή που ζήτησε το Κοινοβούλιο σχετικά με τις ε, πρωτοβουλίες ε, Ευρωπαίων πολιτών και περιμένουμε και τα πορίσματα της τελικής μελέτης που θα καλύψουν το σύνολο του κύκλου. καθότι θα υπάρχει τουλάχιστον μία πρωτοβουλία πολιτών, ίσως και περισσότερες μέχρι τότε, προς τις οποίες θα έχει ανταποκριθεί η Κομισιόν, καθότι οι διοργανωτές δηλώνουν ότι έχουν συλλέξει περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές και αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία της εξακρίβωσης. Αυτές θα υποβληθούν στην Κομισιόν πολύ σύντομα. Επίσης ε, και άλλες πρωτοβουλίες αυτού του είδους είναι πολύ θετικές όπως το ερωτηματολόγιο το οποίο διοργανώνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής γιατί τα διάφορα αυτά βήματα θα βοηθήσουν σε μια πληρέστερη εξέταση των πρωτοβουλίων πολιτών και εν ευθέτω χρόνο όπως προβλέπετε στον κανονισμό για τις πρωτοβουλίες. Η Κομισιόν θα προετοιμάσει την έκθεσή της μέχρι τον Απρίλιο του 2015 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αυτή. Προς το παρόν η Κομισιόν θεωρεί ότι, ότι είναι ένα πολύ πρόσφατο μέσο οι πρωτοβουλίες πολιτών. Είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε την εφαρμογή τους, όμως ήδη έχει σημειώσει κάποιες πρώτες επιτυχίες. Από τις πρώτες δέκα καταχωρισμένες πρωτοβουλίες υπάρχουν τρεις που δηλώνουν ότι έχουν φτάσει τα απαραίτητα όρια του ενός εκατομμυρίου υπογραφών και των συμμετοχών από κράτη-μέλη. Το οποίο σημαίνει ότι συνολικά Υπάρχουν άνω των 5 εκατομμυρίων δηλώσεις στήριξης που έχουν υπογραφεί από Ευρωπαίους πολίτες σε όλο το έδαφος της Ένωσης, το, το οποίο μας δείχνει σαφώς ότι αυτό το μέσο έχει αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστό. αυτή τη στιγμή διεξάγονται και ενθαρρύνεται να διεξάγονται συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη και παρότι δεν είναι πάντοτε οι προσπάθειε επιτυχής ω προ τη συλλογή του ενό εκατομμυρίου υπογραφών, οπωσδήποτε αυτό βοηθά να οικοδομηθεί ένα υπερεθνικός διάλογο για ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνον τώρα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το πόρισμα αυτό της μελέτης αυτής και ίσως είναι ακατάλληλη χρονική στιγμή να απαντήσω σε όλα τα ζητήματα που φύγονται θα ήταν υπερβολικά λεπτομέρειες κάτι τέτοιο. Τέσσερα επιμέρους σημεία ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς τα μέλη της Επιτροπής που πρέπει να προέρχονται από 7 διαφορετικά κράτη-μέλη είναι μια πολύ καλή ιδέα πιστεύουμε ότι υφίστανται πλατφόρμες που βοηθούν την επαφή μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών από διάφορες χώρες και την αναζήτηση εταίρων για τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας, διότι η διοργάνωση είναι τεράστιο ζήτημα απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και η συμμετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα στην Οργανωτική Επιτροπή, είναι κέρια σημασίας. Και μια πρωτοβουλία ποτέ δεν μπορεί να διοργανώνεται από άλλους φορείς για λογαριασμό εκείνων που θέλουν να προωθήσουν την πρωτοβουλία αυτή και να προχωρήσουν σε αυτήν την εκστρατεία, αν θέλετε, αναζήτησης στήριξης. Έχουν ακουστεί και επικρίσεις σχετικά με την απέτηση αυτή των 7 διαφορετικών κρατών μελών και ήταν λίγο ανησυχητικό να βλέπει κανείς ότι αφενός είναι δύσκολο να βρει κανείς τους ανθρώπους, τους πολίτες που θα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια τόσο εντατική προσπάθεια επί 12 μήνες, αλλά είναι προϋπόθεση. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μια επιτροπή θα μπορούσε να συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές, εφόσον οι πολίτες που έχουν καλές ιδέες δεν καταφέρουν να βρουν εταίρους συνεργασίες στα άλλα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διοργανώνονται επαφές, δίκτυα, πλατφόρμες, αλλά αυτή η προαπέτηση της Οργανωτικής ε, Επιτροπής με 7 πολίτες από 7 διαφορετικά κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντική και δίνει και την, ε, αν θέλετε, δυνατότητα να είναι επιτυχής μια τέτοια προσπάθεια και στην επόμενη φάση, στο επόμενο στάδιο να αναφερθώ τώρα στην χρηματοδότηση. Δεν, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω δει ποτέ το μέγεθος του ενός εκατομμυρίου ευρώ. σχετικά με την ε, διαχείριση της πρωτοβουλίας. Τώρα δεν έχω μπροστά μου και δεν θυμάμαι απ' έξω τα μεγέθη, αλλά νομίζω ότι τα μεγέθη αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας για το δικαίωμα στο νερό νομίζω ότι είναι 100.000 ευρώ ή ίσως υπάρχουν και κάποια πρόσθετα μεγέθη. Δηλαδή ίσως το τελικό μέγεθος να είναι 160.000 αλλά εν πάση περιπτώσει η τάξη μεγέθους που θυμάμαι είναι αυτή για την πρώτη επιτυχή πρωτοβουλία είναι προφανής ότι όσο, όσο περισσότερους πόρους έχει κανείς διάθεσή του τόσο ευρύτερη εκστρατεία μπορεί να διεξαγάγει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι προαπέτηση το 1 εκατομμύριο ευρώ για τη διεξαγωγή μιας ICI. Ιδιαίτερα με την προσφορά της Κομισιόν να φιλοξενεί τη συλλογή, τη διαδικτυακή συλλογή της υπογραφής για την οποία δεν επιβαρύνονται οι διοργανωτές Επίσης η εξακρίβωση των υπογραφών δεν επιβαρύνει τους γεωργαντές. Και τι άλλο σημείωσε. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί πραγματικά είναι η πρώτη φορά που βλέπω τη μελέτη αυτή, λέει ο μιλήτρια. Τα κοινωνικά μέσα κάθε αυτά επίσης δεν επιβαρύνουν. Αυτό που επιβαρύνει είναι η ίδια η εκστρατεία. Και επίσης ήθελα να αναφερθώ στους κανόνες σχετικά με τις υπογραφές. Στην πρόταση κανονισμού της Κομισιόν είχαμε έναν ενιαίο μορφότυπο με ίδιες προαπαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα που θα πρέπει να υποβάλλονται από τους πολίτες. κατά την υπογραφή δήλωσης στήριξης μιας πρωτοβουλίας. Αυτό τροποποιήθηκε με νομοθετική διαδικασία κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου και αυτή τη στιγμή ο κανονισμός λέγει ότι οι προαπαιτήσεις δεδομένων που θα πρέπει να υποβάλλονται καθορίζονται σε κάθε, για κάθε διαφορετική περίπτωση και για κάθε διαφορετικό κράτος μέλος. Αυτό έχει το ατυχές αποτέλεσμα κάποια κράτη-μέλη να ορίζουν τα δεδομένα αυτά σε σχέση με τους υπηκόους τους, για παράδειγμα τον αριθμό εγγράφου ταυτότητος, που μπορεί να υπάρχει μόνο για τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας βεβαίως. Και, αυτά δεν αφορούν τους κατοίκους που όμως δεν είναι υπήκοοι. Εφόσον λοιπόν ένας υπήκοος κράτους μέλους διαμένει στη χώρα του δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως διαμένει σε χώρα που δεν είναι η χώρα της υπηκότητός του και αυτό γίνεται σε διάφορες, διάφορους συνδυασμούς μεταξύ χώρας υπηκότητος και χώρας διαμονής και στο πλαίσιο των κανόνων αυτών μπορεί ή δεν μπορεί ένας τέτοιος πολίτης που ανήκει σε μία από αυτές τις κατηγορίες να δηλώσει ή όχι υποστήριξη προς μία ICI. Η Κομισιόν λοιπόν συστήνει ζωηρά στα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν τους κανόνες αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την μελέτη σχέδιο εκθέσεως. Χαίρομαι που τη ζητήσαμε τη μελέτη αυτή και χαίρομαι που βλέπουμε τα πρώτα ευρήματά σας. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλό και χρήσιμο το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας από το... την αρχή που αναλάβατε μέχρι τώρα. Βλέπω, και δεν ήταν πολύ ο χρόνος, να έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πολλή δουλειά, πολύ χρήσιμο και νομίζω ότι και εκ μέρους της Επιτροπής μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι απολύτως απαραίτητο να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο δημιουργήσαμε με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δεν έχει προηγούμενό του στον κόσμο. Είναι η πρώτη φορά που θεσπίζεται ένα διεθνικό μέσον συμμετοχής των πολιτών, άρα δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, άρα πρέπει να μάθουμε όσο προχωράει, άρα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί και να βελτιώσουμε το μέσον αυτό καθοδόν. Εξού και είναι πολύ χρήσιμη αυτή η μελέτη γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια, κάποια προβλήματα και πρέπει να τα επιλύσουμε να, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Και αποφασίσαμε το 2015 να γίνει η αναθεώρηση του συστήματος Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας των Πολιτών. όλα αυτά που μας λέτε θα είναι πολύ χρήσιμα για την αναθεώρηση. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που θα μπορούσαν ενδεχομένω αμέσως να εφαρμοστούν. Παράδειγμα, αναφερθήκατε και από την Επιτροπή για τις προϋποθέσεις ε, να υπογράψει κανεί μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Επιτροπή θα ήθελε ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπω άλλωστε και εμεί και συζητήσαμε τι χρειάζεται. Ρωτήσαμε και τα κράτη-μέλη να μα πούνε τι προποθέσει ορίζουν για την επαλήθευση τη υπογραφή και θα ήταν δυνατόν όντω να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ε, φορμάτ, ένας ευρωπαϊκός μορφότυπος και παρόλα αυτά ήρθαν τα κράτη-μέλη στις απαντήσεις τους και μας λέγανε άλλο η Ελλάδα, άλλο η Ρουμανία, άλλο η Ιταλία που μας έλεγε άμα δεν έχουμε έτσι δεν επικυρώνουμε τη διαδικασία. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο ε, διονγκώθηκε υπερβολικά όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στις εθνικές προϋποθέσεις για το κάθε κράτος χωριστά. Πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκές προϋποθέσεις. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Ξέρετε ότι κάποια στοιχεία των παραρτημάτων 2 και 3 αλλάξαν ήδη το τελευταίο Ιούλιο. Και αν δεν απατώμε, το Λουξεμβούργο είπε δεν απαιτώ αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το διαγράφω αυτό από τις προποθέσεις μου. Ενώ την ίδια στιγμή η Ισπανία έλεγε εγώ θέλω, απαιτώ αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Και το προσέθεσε στις προποθέσεις της. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει «Α, είμαι Ευρωπαίος πολίτης και υπογράφω» πρώτα πρέπει να πει ποια είναι η ηθαγένειά του, τι διαβατήριο έχει, Γάλλος, Ισπανός και αναλόγως και οι υποθέσεις για την ε, υπογραφή. Αυτό είναι το και σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που έχουμε και για το λογισμικό ακόμη, γιατί είναι τόσο περίπλοκο το σύστημα. Μπαίνει κανείς ως Ρουμάνος πολίτης, παραδείγματι, και ανοίγει ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο καταχώρησης από ό,τι για τον Βρετανό πολίτη Φερρυπίν. Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα και οπωσδήποτε με την αναθεώρηση πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο. Δεν μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε εάν δεν συνεργαστούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο τα κράτη-μέλη. Αυτό ήδη μπορούν να το κάνουν από τώρα. Και άπαξ και βρεθεί αυτή η λύση μπορούμε με κάτι εξουσιοδότηση πράξη να υλοποιήσουμε τις τροποποίησεις και αυτήν και άλλες από προβλήματα που έχουμε ήδη εντοπίσει. Γιατί υπάρχει και άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα ήταν να επιτραπεί σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να ξεκινήσει μόνη, να ορίσει μόνη της ποια είναι η αφετηρία της. Το 12 μήνο πολλοί σας είπαν ότι ε, δεν αρκεί. Προβλέπεται όμως από τον κανονισμό. Έστω. Εφόσον προβλέπεται από τον κανονισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πολίτης μπορεί να ξεκινάει μια πρωτοβουλία την 1η Ιουλίου και να έχει 12 μήνες μπροστά του. Αλλά δεν μπορεί να το ορίσει ο μόνος του. Τον ενημερώνει η Επιτροπή. Και με το που θα του δώσει η Επιτροπή το πράσινο φως αμέσω πρέπει να αρχίσει να τρέχει, ενώ δεν είναι ενδεχομένω έτοιμο, δεν έχει το σχετικό υλικό, το έντυπο, δεν έχει αναπτύξει την επικοινωνιακή του πολιτική, δεν έχει μπορέσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μέσων μαζική ενημέρωση, όλα αυτά που χρειάζονται. Αυτά λοιπόν με κάποιε μικρέ αλλαγέ πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την ε, πρωτοβουλία. Αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω ότι μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο συντάξατε την έκθεσή σας, η ανάλυση, το πλαίσιο, πώς λειτουργεί, τα προσκόμματα και εν τέλει προτινόμενες λύσεις. Και αυτό νομίζω ιδιαίτερα για τους ευρωβουλευτές, γιατί βέβαια ε, ίσως να μην μπορεί ο καθής να διαβάσει ολόκληρη την έκθεση, αλλά όταν κανείς θέλει να δει τι είδους εμπόδια εντοπίζονται και τι είδους λύσεις προτείνεται, ε, τότε ναι, μπορούμε να τα συζητήσουμε νομίζω πολύ πιο εύκολα με αυτή τη βάση του εγγράφου σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη δουλειά σας, τη δουλειά που ξεκινήσατε. Σας εύχομαι. Να έχετε την καλύτερη δυνατή έμπνευση, ενημέρωση και αρρωγή από κάθε πλευρά και εύχομαι κάθε επιτυχία για την έκθεση και την περαιτέρω δουλειά πάνω σε αυτή την έκθεση, τη μελέτη. Θα περιμένουμε να δούμε και τα οριστικά αποτελέσματα και να Ξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Χουντή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Παρακολούθησα το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης της έκθεσης και θέλω να ευχαριστήσω. Σύντομα παρατηρήσεις με τι οποίε στιγμή που γράφτηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας αυτή η τι ενισχυω απο τη στιγμη που γραφτηκε στη συνθηκη της λισαβονας αυτη η δυνατοτητα μέχρι τα σήμερα, η πρώτη διαπίστωση είναι ότι δεν είναι πολύ γνωστή ή δεν είναι τόσο γνωστή ούτω ώστε να κινητοποιηθούν οι πολίτε. Μια πρώτη διαπίστωση. Στη χώρα μου, παραδείγματο χάρη στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει το νερό. Επομένω, χρειάζεται μια εκστρατεία ε, για να γίνει γνωστή αυτή η δυνατότητα. Και μιλώ πολύ πρακτικά. Αυτή η εκστρατεία γνωστοποίηση των δυνατοτήτων μπορούν να γίνουν από διάφορου φορεί ας πούμε από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε χώρα, από τις αντιπροσωπείες της Κομισιόν σε κάθε χώρα, που έχουν και τις τεχνικές δυνατότητες στις ιστοσελίδες τους, σε άλλα site, πέρα από τις προσπάθειες που μπορεί να κάνει κάποιος με δική του πρωτοβουλία. Επομένως, αυτή η εκστρατεία για να γίνει γνωστή αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να κλιμακωθεί. Το δεύτερο, με βάση την έκθεση, αλλά και όταν κουβεντιάζονταν ο κανονισμός, έγινε νομίζω φανερό ότι ενώ είναι μια πρωτοβουλία που έχει αυτές τις δυσκολίες να γίνει γνωστή, να συλλεγούν κτλ. Όταν οι δυσκολίες είναι χρονοβόρες και έντονα γραφειοκρατικές, ουσιαστικά την ακυρώνουν αυτή την πρωτοβουλία, καθώς για ένα θέμα που μπορείς να συγκεντρώσεις ένα τέτοιο αριθμό, ίσως έχει φύγει από την επικαιρότητα ή έχουν προκύψει κάποιες αλλαγές που κάνουν τον πολίτη να μην τη βλέπει ως κάτι το άμεσο. Προφανώς είναι συσσωρευμένα κάποια προβλήματα και μπορεί να πει κανείς είμαστε έτοιμοι για κάτι. Αλλά στη συνέχεια της και για την χρησιμότητα πρέπει μια σειρά δυσκολίες που εντοπίστηκαν και άλλες που μπορεί να κανείς να εντοπίσει πρέπει να διορθωθούν για να μπορέσει να συνδεθεί το άμεσο και το επίγον του ζητήματος που θέτει η πρωτοβουλία με την τελική της υλοποίηση. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, γραφειοκρατικές διαδικασίες και χρονοβόρες δυσκολίες το κάνουν να χάνει το ενδιαφέρον του το θέμα. Κατά τη γνώμη μου ως πολύ γενική παρατήρηση. Και το τρίτο, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και την εκπρόσωπο της Κομισιόν. <clears throat> Αν δεν δει ο πολίτης, έστω πιλωτικά, το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, δεν θα μπορέσει αυτό το πράγμα να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στο μέλλον. Να το κάνω πιο απλά, πιο απλό και είναι κατανοητό. Αυτή η πρωτοβουλία είναι νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών από τα κάτω. Δεν είναι δεσμευτική για την Κομισιόν και εδώ το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την ευαισθησία που θα δείξει και επιτρέψτε μου να πω και από τη γρηγοράδα που θα δείξει. Έστω και για την, πρώτο, την πρώτη πρωτοβουλία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Ότι η Κομισιόν, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν μια ευαισθησία και με την πρόταση που διατυπώθηκε έφτιαξαν μια έκθεση για να συζητηθεί επί της ουσίας το θέμα με τις προτάσεις που έγινε. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις και ευχαριστώ και πάλι για την έκθεση γιατί μας δίνει πάρα πολλές ε, σκέψεις, ε, ναι, πάρα σκέψεις για να βελτιωθούν μια σειρά πράγματα και να μπορέσει να αξιοποιηθεί προ όφελο των πολιτών μια αυτή πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Συνεπώς μπορούμε να κλείσουμε με το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις μελέτες σας, για την παρουσία σας εδώ και την παρουσίασή σας. Θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερος χρήσιμη. Ξέρετε ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε την πρώτη ακρόαση γύρω από τα θέματα αυτά και γι' αυτό η, τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν και οι προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στη μελέτη σας θα ληφθούν υπόψη και φυσικά και θα εφαρμοστούν. Βέβαια η έκθεση αυτή είναι η ενδιάμεση έκθεση και θα συνεχίσουμε περιμένοντας την τελική διατύπωση. Ελπίζω στο μέλλον να συνεργαστούμε καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της ε, εφαρμογής της πρωτοβουλίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τα μέλη που πήραν το λόγο, τέλος της συνεδρίασης.